I would like to start the meeting because... Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνεδρίαση, γιατί περνάει ο χρόνος γρήγορα. Σας καλωσορίζω όλους. Ξεκινώ με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης. Και σας ενημερώνω ότι, ως συνήθως, έχουμε μετάδοση από διαδίκτυο τη συνεδρίασης. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη έγκριση. Σας έχει διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη. Μία τροποποίηση έχω να σας προτείνω για την αυριανή συνεδρίαση, γιατί στο σημείο 8 του σχεδίου έχουμε αύριο συνεδρίαση με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Φραν Τίμερμανς ο οποίος δυστυχώς θα πρέπει να μεταβεί κατεπηγόντως στην Ιταλία. Σχέση με το πρόβλημα των προσφύγων, δεν θα μπορέσει να έρθει λοιπόν σε εμάς. Αύριο θα αρχίσει τις 10 συνεδρίαση. θα σας ε, έρθει και η ενημέρωση από, το, από τη γραμματεία μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ότι αρχίζουμε στις 10 αύριο. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αλλαγές, κάνουμε την τροποποίηση και εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και πάω στο επόμενο σημείο που είναι οι ανακοινώσει της Πρόεδρου. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση με την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα θυμάστε πως είχαν προτείνει οι να έρθουν εδώ. Ναι, και έρχονται πότε πότε στις Βρυξέλλες. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 1.30 με 3 το απόγευμα, στην αίθουσα ASP 5Ε2 ε συνεδρίαση με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχετε ενημερωθεί από τη Γραμματεία. Οι πολιτικέ ομάδε έχουν αποστείλει τη σχετική ενημέρωση για του συναδέλφους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, αλλά βέβαια όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Η συνεδρία δεν λαμβάνει χώρα στη συνήθεια ώρα διεξαγωγή των συνεδριάσεών μα Είναι πάντω ανοιχτή προ όλου του βουλευτέ. αν δεν απατώμε. Η συνεδρίαση αυτή, όποιος από το Κοινοβούλιο θέλει να έρθει, είναι ευπρόσδεκτο. Η μόνη δυσκολία είναι ότι δεν έχουμε διερμηνία. Θα γίνει μόνο στα αγγλικά η συζήτηση. και ζητώ συγγνώμη από όποιον από εσά ε, δυσκολευτεί και δεν μπορέσει να παρευρεθεί λόγω αυτού του ζητήματο τη γλώσσα. Στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη, υπαριθμών 3. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο εισηγητέ, ο Ιωλάινεν και υποφαινομένοι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τι τροπολογίε που μας ε, αποστήλατε. Έχουμε τροπολογίες και για το σχέδιο εκθέσεως και για το ψήφισμα. 284 για το σχέδιο εκθέσεως. Συνολικά. Και 76 για την εκλογική πράξη 208 για το νομοθετικό ψήφισμα. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με το γιο, συναντήσαμε τους σκιώδεις, σε μια συνεδρία συναντήσαμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους και να βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις αυτή την εβδομάδα και θέλω να σας ενημερώσω ότι σκοπεύουμε την ψηφοφορία Τη έκθεση να την προβλέψουμε για την 28 Σεπτεμβρίου, προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Έτσι ώστε στην ε, σύνοδο του Οκτωβρίου να υποβληθεί το θέμα στην έγκριση της Ολομέλειας. Ίσως να θυμάστε, πάντως δεν θέλω να σας ενημερώσω ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε έγκυται στο γεγονός ότι το στο Συμβούλιο απαιτείται ομοφωνία και στο Συμβούλιο η διαδικασία για την έγκριση περνάει και από τις εθνικές κυρώσεις, από τις εθνικές αναμεστάξεις. Έτσι, στη διατύπωση των τροπολογιών της εκλογικής πράξης του 1976 προσπαθούμε να λαμβάνουμε υπόψη και αυτές τις προκλήσεις. Γιατί από τις επαφές μας με το Συμβούλιο αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη πρόκληση. Η ιδέα μιας ε, διεθνούς λίστας ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο, προκειμένου να εξετάσει αυτή τη ε, μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο, απαιτεί να μην υπάρξει αυτή η πρόταση στο Κοινοβούλιο. Και βέβαια όταν πρόκειται για εκλογική διαδικασία πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί στο τι μπορούμε να επιτύχουμε. Κάποιες λοιπόν παραχωρήσει από το Συμβούλιο μπορούμε να τι εξασφαλίσουμε, αλλά με τις ε, δεδομένες πολιτικές ε, ισορροπίες κάποιες λύσεις δεν μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε. Αυτό θέλω να σα ενημερώσω. Γιώ, θέλεις να λάβεις το λόγο τώρα και να επανέλθω εάν ε, έχει κάτι να συμπληρώσω. Γιώ Λάινεν παρακαλώ. Το δικό μου το μικρόφωνο δουλεύει και έτσι έχω απόλυτη εξουσία, αλλά είναι κάποιος, κάποιο άλλο μικρόφωνο. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του τεχνικού μας. Α, ωραία, τώρα δουλεύει. Μάλιστα, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βλέπω με χαρά ότι υπάρχει ευρύτατο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, για τις 200 ε, ε, τόσες τροπολογίες. Νομίζω ότι μια σειρά από ζητήματα μπορούν να εξασφαλίσουν ευρύτατη τη συνένεση. Όπως έδειξε και η πρώτη συνεδρία των συντονιστών και των σχεδόν των εισηγητών. Διαφάνεια επιδιώκουμε, δημοκρατικές προδιαγραφές κατά τον προσδιορισμό των υποψηφιοτήτων και των προβεβλημένων υποψηφίων για τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Έτσι ώστε να υπάρχει στον αυτόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ κομμάτων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί βλέπουν ότι πρέπει να βελτιωθεί η ορατότητα για τον πολίτη των ευρωπαϊκών εκλογών. Και ιδιαίτερα σε αυτό υπάρχει ευρύτερη συνένεση ισομερής εκπροσώπηση των φύλων πρέπει να διαφυλαχθεί, σε αυτό συμφωνούμε. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρκετά κράτη χρειάζεται να εξασφαλιστεί πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Θα δούμε λοιπόν ποια διατύπωση θα κρυθεί ως η καλύτερη. Έχουμε επίσης νομίζω συνένεση ως προς ε, περιορισμένες εμβέλειας ζητήματα για την κατάθεση φερρυπίν για την προθεσμία κατάθεση των υποψηφιωτήτων, των καταλόγων των υποψηφίων και ω προ το ζήτημα ότι δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται αποτελέσματα μέχρι ότου κλείσουν όλα τα εκλογικά κέντρα. Αυτό θα ισχύει για όλα τα κράτη. Κάποια ζητήματα έχουμε ακόμα να επιλύσουμε, να συζητήσουμε. Το ελάχιστο όριο για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3 έως 5%. Ένα από τα ζητήματα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να ε, μας απασχολεί στο ζήτημα της λειτουργικότητας του Κοινοβουλίου. Και βέβαια στο θέμα της ε, ισότητας των ευκαιριών σε κάθε, κάθε επίπεδο πρέπει να προβλεφθεί ένα ελάχιστο όριο κατά 3% τουλάχιστον ε, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή εκπροσώπηση. Αυτά έχω να πω προς το παρόν και περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα ίσως και εγώ να προσθέσω κάτι, δηλαδή ότι γνωρίζουμε όλοι πώς είναι το εθνικό σύστημα και πώς αντιμετωπίζονται οι εθνικές ε, εκλογές και οι ευρωπαϊκές εκλογές και βεβαίως δικό μας στόχος είναι να υπερκεραστούν οι ε, πολιτιστικοί φραγμοί ε, έτσι ώστε να υπάρξει όχι μόνο αλλαγή του εκλογικού νόμου αλλά και αλλαγή της αντίληψης ε, που έχουν οι πολίτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της διασύνδεσης ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να, γίνει, να ισχυροποιηθεί και η, αντίληψη που έχουν οι πολίτες για αυτές τις εκλογές ε, και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ε, φαίνεται να μην είναι πολύ ε, ε, να, να μην γνωρίζουν ακριβώς, ε, να μην δίνουν μάλλον την σημασία που πρέπει στις ευρωπαϊκές εκλογές, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Σέφλινγκ είναι ο πρώτος που θέλει το λόγο. Ωραία, τώρα ακούγομαι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι συζητήσαμε το θέμα αυτό πολλές φορές. Ε, αναφερθήκατε ε, σε ένα σωρό ονόματα που δίνουμε στην ιδέα αυτή, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για μια ιδέα που ακόμα δεν έχει οριμάσει. Εγώ είχα αναμειχθεί στο προηγούμενο κοινοβούλιο, δηλαδή στην προηγούμενη θητεία, ε, με το θέμα αυτό και συνεπέρανα ότι και το ίδιο το Κοινοβούλιο είναι βαθιά μοιρασμένο στο θέμα αυτό κυρίως τα μικρότερα κράτη-μέλη, τα οποία φοβούνται ότι εάν λειτουργήσει αυτή η πανευρωπαϊκή λίστα, τότε αυτά θα περιθωριοποιηθούν, αυτές θα περιθωριοποιηθούν. Είναι ένας φόβος ο οποίος υποβόσκει. Νομίζω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπέρ βέβαια. Ε, τώρα, εάν προκύψει κάτι και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, με επιθυμούν ε, να γίνει κάτι, ε, τότε θα πρέπει να συζητηθεί σε στην περίπτωση της σύγκλησης μιας συνάντησης ε, για την ε, συνθήκη αυτή. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να δοθεί κυρίως το ευρωπαϊκό πρόσημο που λείπει και αυτό είναι, εκεί έγκυται και η δυσκολία. Νομίζω ότι ε, για τους περισσότερους από μας υπάρχει μία κίνηση η οποία τραβάει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές προς τις εθνικές εκλογές. Ε, και προς το εσωτερικό των χωρών. Θα πρέπει να φτάσουμε στη φάση κατά την οποία οι ευρωπαϊκές εκλογές θα γίνουν πραγματικά ευρωπαϊκές ε, και νομίζω ότι εκεί έγκυται και η δυσκολία η αλλαγή στο σύστημα θα πρέπει να δημιουργήσει, να δώσει περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα στις εκλογές και τότε θα είμαστε σε καλό δρόμο. Ε, ξέρετε, προσωπικά, οποτεδήποτε μιλάω, ας πούμε, ε, στην Ουγγαρία για τις ευρωπαϊκές εκλογές ε, και όλοι ανοίγουν διάπλατα τα μάτια τους από έκπληση και λένε ό, αυτό δεν το ξέραμε, α, τι μου λες, έτσι είναι». Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωριστούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές από τις εθνικές πολιτικές ε, και τότε θα είμαστε στον καλό δρόμο. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε ελάχιστο κατόφλι. Νομίζω ότι ακούσαμε ε, τα επιχειρήματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και επιθυμητό θα έλεγα εγώ, ευκταίο, να υπάρχει ομοιομορφία ε, στις 28 χώρες ε, γιατί στο τέλος τέλος μιλάμε και για ένα κοινοβούλιο, ενιαίο κοινοβούλιο και επομένως αυτό θα πρέπει να καθορίσει τους κανόνες ε, που θα το διέπουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εσά ε, ε, είπε για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και τον τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Είχα την αίσθηση ότι ακόμα είναι ανοιχτό το ζήτημα της ε, διεξαγωγής των εκλογών, είναι εθνικό θέμα, αλλά πάντως ε, τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από κοινού την ίδια στιγμή, μάλλον Κυριακή βράδυ. Αλλά ε, ε, ε, θα ήθελα αυτή την ερώτηση να κάνω σχετικά με την ώρα και μέρα διεξαγωγής των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ, Μόρτεν Μέσο Σμιτ. Πρέπει να πατήξω σωστή τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Τέλος πάντων. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με όσα είπε ο Τζόρς, ότι είναι άκρος ε, αυτή η έκθεση. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι ελπίζω δεν να μην φτάσουμε και ποτέ σε αυτό το σημείο όπου δεν θα θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι έχουν καμιά ε, διαφορά μεταξύ τους, γιατί είναι ένας και μόνο λαός. Εάν η ψηφοφόροι μου, έστω και ένας, έβλεπε, που δεν το θεωρώ και πιθανό αυτή την ε, συνεδρίαση, θα άκουγαν μία ε, φωνή και μόνο, τη φωνή του διερμηνέα αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μία ε, φωνή εδώ σε αυτό το κοινόβουλο που στα αγγλικά και στα γαλλικά ε, προέρχεται από το ρήμα μιλώ, παρλάρε. Το θέμα είναι η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό είναι και τόσο ωραία η δημοκρατία και γιατί υπάρχει το κράτος δικαίου και για τα θεσμικά όργανα. Και ελπίζω αυτό να επικρατήσει σε όλη την Ευρώπη. Όμως ε, αυτό το θεσμικό όργανο έχει μία δομή από πάνω προς τα κάτω. Δεν ε, υπάρχει αυτό όμως στο DNA του κόσμου και πιστεύω ότι είναι επιβλαβές και η έκθεση αυτή είναι επιβλαβής γιατί η δημοκρατία, παραβιάζει την αρχή της γι' αυτό και θα πρέπει η ομάδα ECR να το απορρίψει και θα το απορρίψει σε μεγάλη πλειοψηφία. Will correct your... Είπατε ότι είναι πρόωρο για τους διακρατικούς καταλόγους αποκλειστικά νομίζω ε, αυτό αφορούσε το σχόλιο ο Τζόρτζ. Ναι, ήταν κάπως σαν πολιτιστική ιδιοποίηση ή απαλωτρίωση, αν μπορώ να το πω έτσι. Η Μετσέδες Μπρέσο. Dovrebbe <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη αφορά το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών. Άκουσα ότι είστε διατεθειμένοι στις τροπολογίες να ε, ε, λάβετε υπόψη μια τροπολογία κατά αυτήν την έννοια που θα μπορούσε να είναι γενικής φύσεως και επομένω ε, να μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες εδώ μέσα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι ελεκλογικοί νόμοι να διασφαλίζουν την ισότητα των γυναικών προσαρμοζόμενοι στους εθνικούς εκλογικούς νόμους κατά περίπτωση. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται περισσότερη όθηση κατά την άποψή μου είναι το θέμα των πληροφοριών που αφορούν ε, τα εθνικά κόμματα και τις ε, ε, τις συμμετοχές αυτών των κομμάτων. Ίσως θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω, όχι μόνο να ενθαρρύνουμε, να πούμε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ήδη το γεγονός ότι στους εκλογικούς, ε, κατα... στους εκλογικούς ε, καταλόγους, ε, στις εκλογικές λίστες μάλλον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν, αυτό είναι ήδη κάτι πολύ καλό. Έχω και άλλη μία παρατήρηση η οποία έκλεισε το μικρόφωνο της κυρίας Μπρέσο. Φαίνεται ότι το μικρόφωνο μου έχει κάποια προβλήματα, ένα βοσβήνει. Εν πάση περιπτώσει, είχα μια συνάντηση με εθνικούς βουλευτές των κάτω χωρών και προέκυψε από τη συνάντηση αυτή ότι θεωρούν ότι η πιο χαμηλή συμμετοχή ε, σε ευρωπαϊκές εκλογές σε σχέση με τις εθνικές εκλογές συνήθως αυτό συμβαίνει αλλά δεν είναι και νόμος ότι αυτό ε, λένε ε, σημαίνει ότι έχουν λιγότερη ας πούμε δημοκρατική νομιμοποίηση οι Ευρωπαίοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω εάν αυτό θα μπορέσει να φανεί κατά κάποιο τρόπο στον εκλογικό νόμο. Αυτό το πρόβλημα, λέω, είναι η ελλειπής πληροφόρηση ε, περί τις ευρωπαϊκές εκλογές και δεν ε, αναφέρομαι μόνο στην έλλειψη των ε, μέσων ενημέρωσης. Όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα μέσω ε, των δημοσίων μέσων ε, μέσα από τρόπους δημόσιας επικοινωνίας, τηλεοράσεις κλπ. Ε, να κοινοποιήσουν κάποια ζητήματα όσον αφορά την πολιτική, τις πολιτικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ελπίς λοιπόν πληροφόρηση περί τις ευρωπαϊκές εκλογές από πλευράς των κρατών μελών. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει συγκεκριμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η ελλειπής γνώση ε, και αντίληψη της ε, ε, ε, σε δημοκρατική νομιμοποίηση που έχουν ε, οι ευρωπαϊκές εκλογές που εκλέγουν μέσα από άμεσες διαδικασίες τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να νομοποιηθεί περισσότερο γιατί το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιο μακρινό και λιγότερο γνωστό στους πολίτες. Νομίζω ότι αν αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την e-δημόκραση ε, θα πρέπει να δουλέψουμε κατά αυτήν την έννοια και προς αυτήν την ε, κάλυψη του κενού, της, ε, του δημοκρατικού ελλείμματος και της ελλειπούς γνώσης των όσων συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο και στις ευρωπαϊκές εκλογές. οι ευρωπαϊκές εκλογές θεωρείται από πολλούς ε, πολίτες από ό,τι φαίνεται λιγότερο δημοκρατική λόγω της μικρότερης συμμετοχής. Βάζω ένα ερωτηματικό, δεν ξέρω εάν γι' αυτό ευθύνεται ο εκλογικός νόμος, αλλά εμείς ως αρμόδια καθήλυν επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι εμπίπτει στις δικές μας ε, ε, ε, αρμοδιότητες αυτό το θέμα της ε, λογοδοσίας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που καθυστέρησα λίγο. Αλλά με ενημέρωσαν για το τι έχει υποθεί μέχρι τώρα. Επανέρχομαι στους διακρατικούς εκλογικούς καταλόγους και καταρχάς θα σας παρακαλέσω να το δούμε έτσι λίγο αυστηρά το ζήτημα είναι το πρώτο ε, κοινοβουλευτικό όργανο και όχι το δεύτερο ε, ενό συστήματο κοινοβουλευτικού με μία άνω και μία κάτω βουλή. Και η συνθήκη λέει, προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ε, υποπίπτουμε σε ένα, ε, σε ένα ασφάλμα λογικής. Μπορεί να πέσουμε και στον τοίχο μπροστά του Συμβουλίου και να γίνουμε σκόνη και αλλά τέλος πάντων δεν είναι τόσο κακό. Αυτή τη συνθήκη την έχουν υπογράψει και επικυρώσει όλοι. Στις ε, επιτροπές σας φαντάζομαι ότι όλοι έχετε προσκούσει το ερώτημα πώς μπορούμε να προασπίσουμε τα ευρωπαϊκά κοινά συμφέροντα. Εκλεγόμαστε σε μια περιφέρεια της Ένωσης ή μπορούμε να νομοθετούμε και τους νόμους ε, να ε, τους ε, αποδέχονται τα 500 εκατομμύρια πολίτες γιατί έχουν συνταχθεί για όλους αυτούς τους πολίτες. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μειοψηφία. Πιστεύω πάντως ότι λάθος κάνει το Συμβούλιο που ενθαρρύνει μια διέρεση, ένα διχασμό εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθεί να χειραγωγήσει κάποιους βουλευτές, αλλά αυτό δεν είναι σωστό αν θέλουμε να έχουμε ποιοτικέ εργασίες και να είμαστε αξιόπιστοι. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω, νομίζω ότι αυτή η έκθεση που είναι το μόνο θετικό κείμενο. Αν ε, αυτό το ζήτημα το διεκπαιρεώσουμε με αυτόν τον τρόπο, παρόλα όσα γράφονται στη συνθήκη, δεν θα μας πει, καμία τιμή και για ε, όλα τα συστήματα που τους αρέσουν πολύ στα πολιτικά κόμματα, δηλαδή μιλάνε για την αρχή της ισότητας, ε, επειδή όμως λένε, ξέρουν ότι ποτέ δεν θα φτάσει μια γυναίκα στα ανώτατα αξιώματα. Ως γυναίκα σας το επισημαίνει και αυτό. Ευχαριστώ. Ακούστε. Εδώ μιλάμε για την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως τουλάχιστον το παρουσίασε ο προηγούμενο ομιλητή. Δεν μιλάμε για την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές εδώ και στην αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αμφισβητήσει σε μια πολύ σημαντική του απόφαση ε, το Σύνταγμα, τη συνθήκη ε, και μιλάω για το Γερμανικό βέβαια Δικαστήριο που δεν είναι και τυχαίο και είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ως κοινότητα αφηρημένη τη ενία, αλλά ως μια κοινότητα που εκφράζεται με εθνικούς τρόπους, κατά κάποιο τρόπο. Υπό την έννοια αυτή, δηλαδή, το ε, συνταγματικό ε, δικαστήριο της Καλσούδης αποφαίνεται ε, αρνητικά σε σχέση με το ζήτημα που μας αφορά και το λέω αυτό γιατί συχνά στη ζωή μας βλέπουμε καταστάσεις όπου Το καλύτερο είναι το εχθρό του, ο του καλού. Δεν θα πρέπει να προτείνουμε λοιπόν τέτοιες λύσεις που θα είναι αντίθετες με τις νομικές παραδόσεις και τις εκλογικές παραδόσεις. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, δεν ψηφίζουν ε, την Κυριακή και έχουν κάθε δικαίωμα να συνεχίσουν να μην ψηφίζουν την Κυριακή. Πολλές και διαφορετικές λύσεις μπορούν και πρέπει να δοθούν και αυτό θα συνιστούσα οι συνάδελφοι να μην σκέφτονται ότι η νομοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι διαφορετικό από το εθνικό πλαίσιο. Αντίθετα θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή τη ε, διαφορετικότητα, το πλούτο, την ποικιλομορφία να την αξιοποιήσουμε και όχι να υιοθετήσουμε μία νέα λύση η οποία θα θα τα εξισώσει όλα. γιατί θα έχουμε ακόμη χαμηλότερη προσέλευση σε ευρωεκλογέ. Ενώ αυτό που θέλουμε είναι να έρθουμε πιο κοντά στο εθνικό πλαίσιο και όχι εμείς να λέμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο από το εθνικό πλαίσιο. Και ε, αναφέρω το σταγματικό δικαστήριο όχι γιατί είμαι υπέρμαχος του γερμανικού δικαστηρίου ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά επειδή συχνά έχω διαφορετικές απόψεις, θα πω από τις ε, απόψεις των Γερμανών πολιτικών εδώ, αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για μια απόφαση, μια ετοιμιγωρία πολύ σημαντική για εμάς, που μας λέει να μην διαχωρίσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο τον πλούτο του εθνικού, των εθνικών διαφορετικών επιπέδων. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Έχω στο παρελθόν εξηγήσει γιατί θεωρώ ότι μια σειρά από προτάσεις δεν είναι οι επιθυμητές ή ευκτές ή εφικτές. Αλλά από αυτά που είπε ο κύριος Μέστερ Σμιτ, οφείλω να σπεύσω να στηρίξω τον εισηγητή. Σε κάποιες από τις παρατηρήσεις του τουλάχιστον. Φαίνεται ότι υπονοείται κύριε Μέστερ Σμιτ ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία όταν επικρατούν διαφορετικές γλώσσες. Τότε πείτε μου, η Ινδία ως δημοκρατία, η η Ελβετία ως δημοκρατικό σύστημα, πώς λειτουργούν. Εμείς συμφωνούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε την διαφορά, την πολιτιστική πολυμορφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις δομές μέσα στις οποίες ε, συνεργαζόμαστε. Πρέπει να βρούμε κοινέ λύσεις κοινά προβλήματα και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πως είναι λογικό να ορίσουμε τους κανόνες εκείνους που δεν θα επιτρέπουν σε κάποιον να ψηφίζει δύο φορές. Ή ας πούμε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οποίο, το οποίο να γνωρίζουν οι πολίτες και να καταγράφεται στο ε, ψηφοδέλτιο. Γιατί πρέπει να το κρύβουμε από τον πολίτη αυτό την ώρα που ψηφίζει. Επίσης, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι υπάρχουν λύσεις για το να μπορεί να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογέ ένας υποψήφιος ε, για επικεφαλής της Επιτροπής. Άρα δεν πρέπει να έχουμε μια έκθεση. Δεν θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να καλύπτονται. Να καταπλήσουν οι τοποθετήσει σα. Η Πρόεδρος. Θα θέλει φαντάζομαι ο κύριος Μέσερ Σμιτ να μιλήσει. Αργότερα όμως. Παρακαλώ. Συμφωνώ πολύ με τα όσα λέει η Σίλβι Γκουλάχ για τις ε, διεθνείς εκλογικές λίστες. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό θα βοηθήσει. Δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Μέσερ Σμιτ, να είμαστε μία χώρα ή να θεωρούμαστε μία χώρα. Η Ευρώπη δεν είναι μία χώρα, αλλά πρέπει να είναι ένα εγχείρημα. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ένα εγχείρημα το οποίο θα προωθούν πολλές χώρες. Οπότε και νομίζω ότι είμαστε μια αφηρημένη κοινωνία, κοινότητα παράδοξο. Ακόμη και να το πούνε οι Γερμανοί αυτό, τι θα σημαίνει μια αφηρημένη κοινότητα, κοινότητα της ουρανής. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι και επιπλέον για το κατόφλι εισόδου στη Βουλή. Αφού φαίνεται να αποτελεί σημείο αναφορά η απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου, θα σα πενθυμίσω ότι έχει απορρίψει το 5% όριο εισόδου στη Βουλή για τη Γερμανία το ίδιο δικαστήριο. Δεν έχει γίνει δεκτό. Άρα εγώ δεν θα συμφωνούσα να υπάρχει όριο. Αν όμως χρειαστεί να καταλήξουμε στη συμφωνία με βάση αυτό, γιατί να μην είναι 3%. Ας είναι 3%, αλλά όχι περισσότερο. Γιατί πάλι ανάλογα με τις εκλογικές περιφέρειες, μπορεί κάποιοι να αποκλειστούν. Και αυτό δεν νομίζω θα βοηθήσει την ε, μεγαλύτερη εγκύτητα και συμμετοχή στην Ευρώπη των πολιτών. Ισότητα των φίλων και ολοκληρώνω για να σας κρατάω. Συμφωνώ με τη Mercedes. Έχω προτείνει και εγώ κάτι ωστόσο, το οποίο είναι συμβατό με αυτό που μας είπε η συνάδελφος. Στη βαθύτερη έννοια της προτάσεως συμφωνούμε. Και μπορούμε πιστεύω να επεξεργαστούμε μια λύση αποδεκτή για την πλειονοψηφία ή και τους πάντες. Ένα-δύο ζητήματα που σχεδόν δεν έχουν συζητηθεί, αλλά είναι σημαντικά. Το όριο της ε, ενηλικίωσης για τον ψηφοφόρο, το 16, το έχει κάνει η Αυστρία, γιατί όχι. Και αν θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στο νέο, να φέρουμε τον πολίτη πιο κοντά στα θεσμικά όργανα, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του, Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό και να φτάσουμε σε ένα κοινό ψήφισμα. Αναπληρωτές ή επιλαχόντες. Αυτός θα αντικαταστήσει τον βουλευτή, αν τυχόν και αρρωστήσει, εν σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, σπάνιες γραμμίζω, αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα του επιλαχόντος ή του αναπληρωτή μάλλον εννοεί ο μιλητής. Είναι σημαντικό για μένα και το, έχουμε το έχω προτείνει εγώ δηλαδή. Μετά τις εκλογές στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο να τοποθετείται για την υποστήριξή του ή την προτίμησή του για έναν ε, υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπής. Μόνο μία προτίμηση θα εκφράσει. Και από εκεί και πέρα το Συμβούλιο ή όπως οργανωθεί αυτό θα κάνει τη δική του πρόταση. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε εκ προημίου την προτίμηση του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό και την ε, παρουσία του, την δυνατότητά του να επηρεάσει τις εξελίξεις, ε, τις εξουσίες του θα ενισχύσει και ταυτόχρονα θα φέρει τον πολίτη πιο κοντά στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ και μετά η Σιλβικουλά. Σας ευχαριστώ. Ε, για αυτά που είπατε και ρωτήσατε κύριε Κόρμπιτ. Ε, και χαίρομαι που έθιξε το θέμα της ε, ε, γλώσσας ε, και μάλιστα άλλωστε, άλλωστε εγώ μιλάω σε αυτόν στη δική του γλώσσα και όχι εκείνος στη δική μου. Εν πάση περιπτώσει το θέμα των τριών γλωσσών είναι εντάξει άλλωστε και είναι οι φερόες που έχουν δικιά τους γλώσσα αλλά δεν το κάνουμε και θέμα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που είπα εγώ είναι ότι η οικοδόμηση της δικαιοσύνης ε, ε, συγγνώμη της δημοκρατίας, ε, δεν μπορεί να γίνει από πάνω προς τα κάτω. Θα πρέπει να γίνει ανάποδα. Και ξέρετε κύριε Κόρμπεν, προερχόμενος από μια χώρα με λαμπρή ιστορία και με καλά λειτουργούσα δημοκρατία, ότι η δημοκρατία προωθείται και προωθήθηκε στη χώρα του από την πίεση και από τη στάση του Βρετανικού λαού. Επομένως, ο κόσμος ε, ε, ζητάει όντως μεγαλύτερο έλεγχο. Ε, δεν νομίζω ότι ε, γίνεται το αντίθετο, δηλαδή ότι αυθόρμητα κατεβαίνει ο κόσμος στο δρόμο και λέει δώστε περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν νομίζω ότι ακόμα και, τα, ακόμα και αυτό που λέτε για τα περίφημα και περιβόητα ευρωπαϊκά κόμματα που θέλετε διακαώς να δημιουργήσετε, δεν είδα να κατεβαίνει ο κόσμο να ξεχύνεται στου δρόμους και να λέει δώστε τους περισσότερες εξουσίες ή βάλτε τους όλου στο κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, οι ιδιαιτερότητε του καθενό, η ιστορία του, το παρελθόν του κτλ. Τούτο βεβαίω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, ε, ε, φυσικά μπορούμε να έχουμε ε, ε, έναν, ε, ένα, μια οδό η οποία θα μας οδηγήσει στην οικοδόμηση αυτού του συστήματος. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1979 είχαμε τους εκπροσώπους των εθνικών χωρών που ερχόταν. Σιλβί. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συζητάμε εδώ. Ξέρετε ότι θαυμάζω τη Γερμανία, αλλά ε, σύμφωνα με την ε, τελευταία απόφαση την, ε, τελικά να γίνεται αναφορά για αυτά που λέτε σε αποφάσεις το, της ε, γερμανικής νομολογίας. Άρα αυτό που δεν θέλουμε θα γίνει. δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι πιο δυνατές θα δίνουν το ρυθμό για ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ θα προτιμούσα να αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει το δικαστήριο της Καλσρούης να ε, ε, υποδεικνύει την θέση του στο Κοινοβούλιο. αυτό που καταλαβαίνω κύριε Μέσοσμιτ είναι ότι σας ενοχλεί αυτή η υπερευρωπαϊκή ευρωπαικη ας πούμε εξουσία αλλά δεν σας πειράζει καθόλου να παίρνετε χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, αμάν πια πρέπει να σταματήσει αυτό. Ε, δηλαδή ε, μόνο όταν ε, όλοι οι ευρωσκεπτικιστές δεν τους αρέσει το ένα και τους ξυνίζει το άλλο, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πληρωθούν, να πάρουν χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούνε και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να έχουμε μια καλή ποιότητα εργασίας εδώ και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι Ευρωπαίοι βουλευτές δεν θα κλείνονται μέσα σε ε, μικρές εθνικές ε, κατηγορίες. Εγώ πιστεύω ότι τα εμπόδια, ακόμα και αν θεωρούνται αναξεπέραστα, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεραστούν, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είμαστε και πολύ μικροί και λίγοι απέναντι στις αναδυόμενες μεγάλες χώρες. Η κυρία Μπρέσο. Όντως, θα πρέπει να σας δώσω μια απάντηση κύριε Μέσο Σμιτ. Ψηφίσαμε τα, τη δεκαετία του 80 ε, τις πρώτες εκλογές ε, και η μόνη χώρα η οποία ζήτησε ε, στους πολίτες της να πούνε εάν θέλουν ομοσπονδιακή Ευρώπη και με 95% πλειοψηφία είπαν ναι με, με μια τρομερή σχεδόν ομοφωνία. ποτέ σε δημοψήφισμα δεν ε, ρωτήσαμε εάν οι χώρες μας ε, θέλουν, ας πούμε, τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, ε, μια ενωμένη φεντεραλιστική, ομόσπονδη τέλο πάντων, πολιτική Ευρώπη. more νομίζω ότι αυτό θα, ε, κατά διαστήματα ξέρανε οι πολίτες ότι δίνουν, δίνουμε μεγαλύτερη ε, δύναμη στην οικονομία, στην εσωτερική. Τώρα ξέρω ότι εάν γίνει δημοψήφισμα μερικές χώρες θα απαντήσουν όχι. Αλλά πόσες είναι αυτές. Γιατί όπως λέτε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα στην ε, πραγματικότητα ήταν υπέρ και όχι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν είναι σαφές και δεν είναι σίγουρο. Αν ρωτήσουμε τη σωστή ερώτηση, θέλετε να μείνετε ή θέλετε να φύγετε, σε μια πραγματική ομόσπονδη Ευρώπη, με όλα τα δημοκρατικά σταθμίσματα και αντισταθμίσματα. another form I don't know what uh, we are exactly. Uh, sure. Uh, το θέμα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Δεν είμαστε μία όλο και πιο στενή ένωση, αλλά δεν είμαστε και ούτε συνομοσπονδία ούτε ομοσπονδία. Είμαστε λίγο το λίγο τ' άλλο. Νομίζω ότι πρέπει, οφείλουμε, να συνεχίσουμε γιατί διαφορετικά τι, θα σταματήσουμε και θα διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. μία απόφαση να προχωρήσουμε μόνο σε οικονομικά θέματα. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση. Δεν θέλουν όμως και αυτό ε, ε, ε, οι πολίτες μας δεν θέλουν μόνο αυτό, θέλουν περισσότερη Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Και στην άμυνα και στην πολιτική και στην εξωτερική πολιτική. Εν πάση περιπτώσει θέλουν δηλαδή περισσότερες βελτιώσεις πολιτικής υφής. Θέλουν μια πιο πολιτική ένωση. Οπωσδήποτε τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί σαφές και ποιος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει, ποιος όχι. Και αν είναι αρκετοί αυτοί που συμφωνούν, ε, να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Δεν θα ξέρουμε διαφορετικά δηλαδή τι πιστεύει πραγματικά η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Τέλος πάντων, θα ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή με την έκθεση Μπροκ και υποφαινομένης. συμφωνώ με τη Σιλβί Γκουλάρ ότι χρήσιμη θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή λίστα, αλλά ε, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές ε, μπορούν να υπάρχουν τοπικές περιφερειακές αρχές. Εγώ εκλέγω τον ε, ε, εκπρόσωπο που θα με εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο, τον, τον διαλέγω σε τοπικό επίπεδο. Ε, δεν έπεται ότι θα πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκό Κολέγιο για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των ευρωπαϊκών χωρών Κοιτάξτε, τώρα το πώς θα εκλέγονται και ποιος θα εκλέγει και αν θα είναι σε τοπικό επίπεδο, γιατί όχι, θα τα δούμε όλα αυτά. Αν είναι κάτι καλό για την ιδέα της Ευρώπης, εγώ θα είμαι υπέρ. Αλλά εάν σταματήσουμε ε, άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να μπουν στον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο, τότε δεν θα ήταν και πολύ καλή ιδέα. γιατί όταν μετά το Συμβούλιο πάρει αποφάσεις εμείς δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πολλή δουλειά πριν υποβληθεί η πρόταση. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή και να επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή σε αυτή την πρόταση. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν καλή ιδέα. ας πούμε η συμμετοχή εθνικών ε, ε, κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεντρική σημασία σε σημείο. Είναι πολιτική, η πολιτική εκπροσώπηση είναι σημαντικό πράγμα και πιστεύω ότι αυτού του είδους η εκπροσώπηση, η πολιτική εκπροσώπηση είναι το πρώτο σημείο του οποίου θα πρέπει να επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή συζήτηση. Ευχαριστώ Μαξ Άντερσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι πίσω από πολλές από τις προτάσεις κρύβεται μια αγανάκτηση για το ότι οι ευρωεκλογέ είναι αυτό που οι πολιτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ε, ε, δεύτερης κατηγορίας εκλογές, δηλαδή λιγότερο σημαντικές από τις ε, πραγματικές εκλογές και έχουν και χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό μπορεί να το λύσουμε ε, με αλλαγές στο εκλογικό νόμο. Το θέμα δεν είναι αν είναι ή δεν είναι δεύτερες κατηγορίες εκλογές ή ευρωεκλογές, αλλά ότι είναι μακριά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους πολίτες. Και η έννοια της συνένεσης και του συμβιβασμού, που είναι κάτι πάρα πολύ καλό, ε, έχει ως αποτέλεσμα παρόλα αυτά οι δημοσιογράφοι η πολιτική και η κοινή γνώμη να μην γνωρίζουν ακριβώς ποιο πρεσβεύει τι. Γιατί στι περισσότερε περιπτώσει καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό που μπορούν να το ψηφίσουν οι περισσότεροι. Αυτό όμω κάνει λιγότερο ενδιαφέρουσε τι εκλογέ γιατί όλοι ψηφίζουν το ίδιο ουσιαστικά. Δεν λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, απλά λέω ότι έχει ως ε, συνέπεια την μείωση του ποσοστού συμμετοχής στις ευρωεκλογέ. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο. Σίγουρα έχουμε και να εξετάσουμε πολλοί τροπολογίες. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν είναι όταν ένα ε, μέλος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, βράχει πρόθεσμα να αντικαθίσταται, να υπάρχει ένας αναπληρωτής ε, από τη λίστα. Αν ε, ο εκλεγής ευρωβουλευτής δεν μπορεί για κάποιο διχρονικό διάστημα να εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Επίσης, το θέμα των κατοφλίων. Στον εκλογικό νόμο υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι οι εκλογές θα πρέπει να είναι αναλογικές. Ωστόσο, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν περιφέρειες πολύ μικρές. Νομίζω στη μικρότερη περιφέρεια εκλέγονται μόνο τρεις βουλευτές. Αυτό δημιουργεί όμως πάρα πολύ ψηλά κατόφλια. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις, εύκολες τεχνικές λύσεις που μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιολάινα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ελεύθερες, άμεσες και οικουμενικές. Φέρουν ως εκ τούτου όλα τα κριτήρια εκλογών που διεξαγόνται σε δημοκρατικά καθεστώτα. Η νομοποίηση λοιπόν του Κοινοβουλίου είναι η ίδια με αυτήν των εθνικών κοινο ή περιφερειακών κοινοβουλίων που εκλέγονται με άμεσες ε, ελεύθερες και οικουμενικές εκλογές. Άρα δεν εξαρτάται από την ε, συμμετοχή ή την αποχή 45. Η 55% η νομοποίηση. Αλλά από το γεγονό ότι δεξάγονται άμεσε οικουμενικέ και γενικέ εκλογέ δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα των ευρωσκεπτικιστών ή των αντιευρωπαϊστών που θεωρούν ότι μια εκλογική αναμέτρηση δεύτερη κατηγορία έχει την ίδια δημοκρατική αξία και την ίδια δημοκρατική νομιμοποίηση με κάθε εκλογική αναμέτρηση που δεξάγεται κατά τρόπο άμεσο, ελεύθερο και οικουμενικό. Βεβαίως, οι ευρωεκλογές θα διεξάγονται στην πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη στιγμή που θα μπορούν πέραν των εθνικών προγραμμάτων και ε, εντολών τα ευρωπαϊκά κόμματα να αντιπαραβάλουν τις, εθνικές, τις ευρωπαϊκές τους δηλώσεις ε, και τα προγράμματά τους και τις εντολές. Τώρα προς τα παρόν έχουμε μια ένωση κρατών και λαών. Άρα Εσπαθεί το επιχείρημα που αναφέρατε ότι εκλέγονται και σε επίπεδο κρατών μελών οι βουλευτές, αλλά ταυτόχρονα ελπίζω ότι θα έχουμε και βουλευτές που θα προκύπτουν από την ε, ενιαία εκλογική περιφέρεια με έναν ευρωπαϊκό κατάλογο υποψηφίων, μια ευρωπαϊκή εκλογική λίστα. Ξέρετε ότι εγώ πάντοτε υποστήριζα αυτή την ιδέα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε παρά τι να την εισαγάγουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία μόνο τότε μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της αν υπάρχει δηλαδή ε, εντολή έδρα καλύτερα βουλευτική, πραγματικά ευρωπαϊκή. Προς το παρόν ακολουθούμε μια διαδική προσέγγιση στην έκθεσή μας με, τους, ε, με τις ε, λίστες που είναι δυνατές να υλοποιηθούν για το 2019 την προσεχή εκλογική αναμέτρηση και μια παράλληλη προσέγγιση με τις συστάσεις για τη γενικότερη πορεία των ευρωεκλογών της ε, εκλογικής νομοθεσίας. Θα πρέπει βεβαίω να συζητηθούν όλα αυτά και ίσως θα πρέπει και να αποφασιστεί το ζήτημα μιας ευρωπαϊκής ε, έδρας και λίστας και Ας μην ε, χάνουμε όμως την εστίασή μας. Ήδη θα δυσκολευτούμε πολύ να εξασφαλίσουμε ομόφωνη ε, απόφαση στο Συμβούλιο μετά όσα έχουμε τώρα προτείνει. Ας μην το καταστήσουμε και αδύνατο έχοντας πρόημα και πρόωρα πριν κανείς αρχίσει να σκέφτεται τι θα φέρουν οι εκλογές του 2019 ε, προτάσεις που δεν είναι όριμες ακόμη να υιοθετηθούν. Είπατε ότι δεν υπάρχει ορατότητα για τις ευρωεκλογέ, δεν ενημερώνονται οι πολίτες και ότι όλοι μας στις περιφερειές μας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον σε αυτή την εκλογική εκστρατεία δύο-τριών μηνών που διεξάγεται για τις ευρωεκλογέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια και το βλέπετε σε μια συμβαστική πρόταση που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες. Ότι δηλαδή θα καταγράφεται ο σύνδεσμος μεταξύ Ευρωπαϊκού κόμματος, Εθνικού Κόμματος και της Ευρωπαϊκής του Οικογένειας, όχι μόνο στο ψηφοδέλτιο, αλλά ότι θα υπάρχει και διαφημιστικό υλικό με εκπομπές και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, με διαφημιστικές ταινίες, ενημερωτικές ταινίες που θα υπογραμμίζουν ε, την υπαγωγή σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα του, του αντίστοιχου εθνικού. Και επίσης θα υπάρξει και διακήρυξη κομματική, το λεγόμενο μανιφέστο των πολιτικών οικογενειών, εκεί όπου θα δηλώνουν τι θέλουν, τι επιδιώκουν, τι είδου Ευρώπη προτείνουν στον πολίτη. Γιατί και αυτό πρέπει να καθίσετε γνωστό. Πολλά είναι τα στοιχεία λοιπόν στη δημοκρατία για τα οποία ο πολίτης ξέρει ότι είναι οι λόγοι και γιατί είναι οι λόγοι για τους οποίους ψηφίζει προς τη μία την άλλη κατεύθυνση και αυτά πρέπει να τα ενισχύουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω από τη συνάδελφη ότι έχετε μάλλον παρερμηνεύσει το δικαστήριο, το σταματικό δικαστήριο της Γερμανίας, της Καρσούης δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θέλαν να περιορίσουν τη δράση του Ευρωπαίου πολίτη. Και εγώ το έχω μελετήσει πολύ αυτό. Δεν ήταν στόχος αυτός. Ε, δεν τους νοιάζει πόσα κόμματα έχουμε στο Κοινοβούλιο. είχαν πει εντάξει μπορεί να είναι 68 διαφορετικά κόμματα γιατί να μείνουν 30 ή κάπου εκεί. Δεν τους νοιάζει αυτό. Και σε αυτό συμφωνώ με τον ε, δικαστή Σοπφλίν ότι είμαστε ένα κοινοβούλιο πρέπει να ε, υπαγόμαστε στους ίδιους κανόνες και να επικρατούν οι ίδιες συνθήκες για τον τρόπο της εκλογής μας. Αυτό που θέλω να σχολιάσω όμως, για το είπε ο κύριος Κάπρας και ο κύριος Άνεμανς, στην περίπτωση που κάποιος ασθενεί ή εγκυμονεί, Φερρυπίν, να αναπληρώνεται από κάποιον βουλευτή. Ωραία. Και αυτός από πού θα προέρχεται, ο αναπληρωτής. Κύριε Κάπρας. Μα από το κατάλογο, από, το, από τη λίστα. Ωραία. Και όταν ε, γιατρευτεί ο πρώτος, ε, γεννήσει κτλ. Τι θα γίνει. Α, θα γυρίζει πίσω. Ναι, αυτή είναι η βασική ιδέα, λέει ο κύριος Κάπρας. Αλλά πρέπει να είναι κάποιος επίσης εκλεγμένος από τον λαό. Πρέπει ήδη να περιλαμβάνεται στην, εκλογικό, στην εκλογική λίστα. Α, εντάξει, λέει ο κύριο Λάινεν, ε, καθώ ε, είχαμε πραγματοποιήσει συνομιλίε με εκπροσώπου εθνικών κοινοβουλίων στο παρελθόν που ισχυρίζονταν ότι δεν έχει σημασία Ποιο είναι ο ευρωβουλευτή ε, και πώ έχει εκλεγεί. Αν τυχόν πέσει, χτυπήσει και χρειάζεται ενάρρωση, τότε θα φέρουν αυτοί κάποιον άλλον για το κοινοβούλιο. Καλώ. Κοιτάξτε, αυτό δεν προβλέπεται σε πολλέ χώρε σαν δυνατότητα. Να αναλάβει κανεί προσωρινά καθήκοντα. Ναι, ξέρω ότι προβλέπεται στη Γαλλία, αλλά όχι και στι 28 χώρε. Επομένω, δεν ξέρω αν είναι καλή αυτή η ιδέα. Είμαι μάλλον επιφυλακτικό. Επίσης ξέρω ότι πολλές χώρες εξετάζουν το θέμα της ε, ενηλικίωσης των ψηφοφόρων και η Αυστρία έχει βέβαια χαμηλό όριο το 16, των 16 ετών και άλλες χώρες, δύο-τρεις τουλάχιστον θεωρούν ότι από τα 16 και μετά μπορεί κανείς να καλείται να συμμετέχει στις δημοκρατικές διεργασίες. Αυτό το έχουμε βάλει αλλά είναι ανοιχτό στις προτάσεις μας, δηλαδή μπορεί ο καθένας να αποφασίσει θέλει. Αλλά μακροπρόθεσμα στα 5-10 χρόνια μπροστά μα. Ξέρετε, οι νέοι στη δεκαετία των 16 ταξιδεύουν, ε, έχουν επικοινωνία με ολόκληρο τον κόσμο. Θα πέσει το όριο αυτό από το 18 στο 16. Ξέρετε, όταν άρχισα εγώ, πρώτη φορά ψήφισα, ήταν ακόμα 21 έτσι ηλικία στο όριο για την ενηλικίωση και κανείς δεν διανοούνταν να το πάει στο 16. Εγώ βεβαίως, καθώς σκέφτομαι και σαν νεαρός, είμαι υπέρ του των 16. Για τον κύριο Τερικαπράς συμφωνώ ότι θα ψηφίσουν οι πολίτες για έναν επικεφαλής υποψήφιο επικεφαλής επιτροπής και μετά θα πρέπει το κοινοβούλιο να ε, ψηφίσει και να ορίσει την πρότασή του για τη θέση αυτή. Αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να οριστεί κάτι τέτοιο στον εκλογικό νόμο, στην εκλογική νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο ξέρετε ότι έχει κατάφερε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση να συναντηθεί με τους υποψηφίου ε, πρόεδρο τη Επιτροπή Δευτέρα και την Τρίτη συνεδρία στο Συμβούλιο. Ε, ίσως να τα καταφέρουμε και την επόμενη φορά. Δεν χρειάζεται να μπει στον εκλογικό νόμο. Μπορούμε να δούμε ποιο έχει τι πλειοψηφίε, ποιον υποστηρίζουμε, ποιον προτείνουμε. Και άρα μπορεί με δυστημία με ένα και ε, διαμαρτυρώμενο για τι όλο και αυξανόμενε ε, εξουσίες του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο να επικυρώσει αυτήν ακριβώ την προτίμησή μα. Η πρόεδρο. Σας ευχαριστώ να προσθέσω και εγώ δύο-τρία πράγματα που σας άκουσα. Να διευκρινίσω ότι σε ό,τι αφορά την απόφαση για την ημερομηνία διεξαλλογής των εκλογών, εμείς προτείναμε με τον Γιώ να, να παραμείνει το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή το κοινοβούλιο να αποφασίζει Υπήρξε πρόταση να είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου πάντα αυτή στην οποία θα διεξάγονται ευρωεκλογέ. Θα δούμε αν θα περάσει αυτή η πρόταση, αλλά δεν ε, σημαίνει ότι θα γίνονται μόνο Κυριακή οι εκλογές σε όλες τις χώρες. Ναι, θέλουμε να κάνουμε μια εναρμόνιση, αλλά όχι ότι θα φέρουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα σε αντιπαράθεση με τα εθνικά συστήματα. Απλά ξεκινάμε από ε, το γεγονός ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στις ευρωεκλογέ και νομίζω ότι είναι καθήκον μας να εξηγήσουμε στους ε, πολίτες ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των ευρωεκλογών και του ότι οι εκπρόσωποι τους Ε, θα έχουν ε, ένα ρόλο που αυξάνεται καθότι θα συμμετέχουν σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Και δεν ξέρω αν εσείς ε, που είστε αρκετά χρόνια στο Κοινοβούλιο φαντάζομαι όμως γνωρίζετε ότι η ισχύ στο Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες, πόσο δραματικά έχει αυξηθεί. Άρα ε, έχουμε την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε την εκλογική διαδικασία και τον εκλογικό νόμο για να δημοσιοποιήσουμε και να μεταδώσουμε στο δυνατόν περισσότερο στον κόσμο το πόσο σημαντικό είναι ότι μπορεί κανείς να επηρεάζει την καθημερινή ζωή όντας ευρωβουλευτής. Και αυτό ε, θα το πετύχει αν δείξει τα ευρωπαϊκά κόμματα, τη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών κομμάτων, αν προσπαθήσει ...να δείξει την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Που σε μεγάλο βαθμό βέβαια θα συνεχίσει να σχετίζεται με τις εθνικές παραδόσεις. Απλά κάπως πληρώνουμε κάποια κενά. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ε, διακρατικές λίστες, υπάρχει μια πρόταση τροπολογίας. Όλα αυτά θα τα ψηφίσουμε, επομένω. Εγώ απλά στην αρχή έθεσα ένα ζήτημα που δεν μου αρέσει καθόλου να θέτω βουλευτή, είναι όμως πραγματικότητα. Ότι δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θα συνεχίσουμε, πρέπει να σας πω, να επεξεργαζόμαστε τις συμβαστικές προτάσεις. Ε, Ξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες ε, που θα τεθούν σε ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τις ομονωμένες τροπολογίες. Ε, θα τα δείτε όλα αυτά. Η ψηφοφορία είναι την επόμενη εβδομάδα, στις 28 του μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Προς το παρόν ολοκληρώνουμε με το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, Γιώργη Σέφλινγκ, να ακούσουμε για πρώτη φορά. Ελπίζω να είναι τελευταία που θα τον ακούμε για το θέμα αυτό. Πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσω σε αυτή την Επιτροπή. Πάντως σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το θέμα αυτό σε τούτη την Επιτροπή. Εξαιρετικά σημαντικά τα όσα ακούστηκαν και οπωσδήποτε χρήσιμα. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ και όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Να πω ότι είχαμε και εξαιρετικά ενδιαφέρους ε, ενδιαφέρον υλικό, input και από την κοινωνία των πολιτών η οποία με ενθουσιασμό συζήτησε το θέμα. Και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό όσον αφορά αυτό το εργαλείο της πρωτοβουλίας των πολιτών. Είναι καινοτόμο εργαλείο, υπό προϋποθέσεις ε, παρέχει στους πολίτες ε, την δυνατότητα να ξεκινήσουν με μία νομοθετικού περιεχομένου πρωτοβουλία, πράγματα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τους συμβιβασμούς, τις συμβαστικές λύσεις, ε, είχαμε μία συνάντηση των συντονιστών, ε, κατά διάρκεια της οποίας συμφωνήσαμε επί πολλών σημείων, όχι 100% βέβαια, ωστόσο ε, καταλήξαμε σε κάποιες επικοδομητικές θέσεις, οι οποίες θα μεταφραστούν σε συμβαστικές τροπολογίες. Τώρα, λέγοντας ότι η, η, η Επιτροπή δεν ήταν ε, και τρομερά γρήγορη. Ήταν αργή, ξεκινήσαμε πριν από 3,5 χρόνια με αυτό το εργαλείο. Φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει και την, ε, ε, το, το βάρος αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήρθε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν σε κάποια στιγμή, σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας ε, και είπε ότι είναι πεπισμένος και ικανοποιημένος γιατί από νομικής απόψεως η Κομισιόν έκανε αυτά που έπρεπε να γίνουν αλλά όσον αφορά την αναγνώριση του πολιτικού βάρους και της διασύνδεσης ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, δεν προχώρησαν τα πράγματα καλά. Εν πάση περιπτώσει ε, καταλαβαίνουμε, ε, την, ε, απεικονίζεται μάλλον έτσι η πρόταση αυτή. Η πρότασή μου, η έκθεσή μου και οι τροπολογίες στόχο έχουν να κάνουν λειτουργικό το όλο σύστημα. Έχω ακούσει και επικρίσεις, όχι από την, την Επιτροπή μας ε, και από το Κοινοβούλιο, αλλά από εκπροσώπους ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών, ότι αυτό το εργαλείο είναι νεκρό, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι οι βελτιώσεις που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκθέσεως αυτής, θα οδεύουν ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή το εργαλείο να γίνει να γίνει πιο εύκολο στη χρήση του, να γίνει πιο απλό. Ε, αυτό ήταν άλλωστε και το σημείο των περισσότερων επικρίσεων. Ενδεχομένως αρχή του επόμενου έτους και όχι τέλος του 2015 ε, θα έχουμε από την Κομισιόν κάποιο αποφασιστικό ε, βήμα έτσι ώστε να γίνει βιώσιμη αυτή η πρόταση, αυτό το εργαλείο. Να πω πάντως ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι περισσότερα θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει γνωστό το εργαλείο αυτό, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Θα μου πει κανείς ότι είναι ένα νεαρό στην ηλικία εργαλείο, όντως, αλλά παρόλα αυτά παρόλα αυτά γίνεται γνωστό μέσω των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνονται από ανθρώπους, δηλαδή από αυτούς ε, που κινητοποιούν ε, ε, τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να μαζευτούν αυτό το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Ε, και επίσης είναι δύσκολο γιατί ε, υπάρχουν 28 διαφορετικοί τρόποι για να ταυτοποιηθεί ο υπογράφων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν υπάρχουν και ταυτότητες τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό πολλές φορές, δεν θέλω να το ξανασυζητήσουμε. Το εργαλείο πάντως μπορεί να δουλέψει, ωστόσο η Κομισιόν θα πρέπει να αποδεχτεί την πολιτική καινοτομία της ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας που δίνεται πλέον στους πολίτες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτός είναι ο στόχος όλου του εγχειρήματος και ελπίζω ότι αυτό τελικά θα επιτευχθεί και θα το καταλάβουν και οι απ' έξω. Πρόεδρος. Όπως ξέρεις, ελπίζαμε να μην σε ξανακούσουμε τοποθετήσει για το θέμα αυτό. Χαίρομαι που δεν έχει πια ε, απαγόρευση η παρουσία μου και η ομιλία μου εδώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο από εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κυρία Κάουφμαν, να εκφράσω θερμά ευχαριστίες στον συγκητή μα Πριν πέρασε στις λεπτομέρειες, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ επικοδομητική η συνάντηση με τους και όλες τους Το βλέπουμε άλλωστε και από τις συμβαστικές προτάσεις που έχουν κατεθεί. Οι οποίες εν γέννη επιτυγχάνουν αυτό που ανέφερε ο κύριο Σόπφλιν τώρα. Ότι δηλαδή γίνεται πιο γνωστό το εργαλείο αυτό και στον πολίτη ώστε να ξέρει ότι έχει τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσει μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών την ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε λοιπόν και στο μέλλον καλύτερα. Και για τις ε, τροπολογίες που έχουν δοτεθεί θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις προκαταρκτικές εκτός από τους συναδέλφους ε, να ξαναμελετήσουν τη δυνατότητα να διατηρηθούν οι τροπολογίες ε, στον τρόπο, στη διατύπωση που έχουν τώρα. Ξεκινώ με τη συμβαστική D, όπου βεβαίως Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την γλώσσα του. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Η πολυκλωσία άλλωστε είναι και ένας από τα πλούτη, από τους πλούτους της Ένωσης μας. Καθίσατε και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό το ζήτημα βέβαια σε σχέση με το, εκλογικό, με το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Ωστόσο, η διατύπωση στη συμβαστική D, δέλτα, απαιτεί πέραν του της αναγνώρισης του δικαιώματος για τη χρήση της μητρικής γλώσσας, όλες και υπογραμμίζω όλες οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με μια πρωτοβουλία των πολιτών να ε, καλύπτονται σε όλες τις γλώσσες. Νομίζω ότι αυτό καθιστά αδύνατη την ε, διαδικασία μπορούμε να χαιρόμαστε ιδιαίτερο για το γεγονό ότι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει εκδηλώσει την ε, διαθεσιμότητά της να προσφέρει τις μεταφράσεις, κάτι το οποίο βεβαίως διευκολύνει ιδιαίτερο τους ε, οργανωτές γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή στα πρώτα χρόνια λειτουργία του μέσου της πρωτοβουλία των πολιτών, δηλαδή τη μετάφραση στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν όμως αυτό, και σημειώνω και υπογραμμίζω για άλλη μια φορά ότι γίνεται λόγος για κάθε και όλες άπασες τις δραστηριότητες. Ε, αυτό δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, γιατί θα έχει πολλά πρακτικά ζητήματα, ποιος θα το οργανώνει και βέβαια τελικά ποιος θα πληρώνει το κόστος, ποιος θα καλύπτει το κόστος. Συμβαστική U, ένα σημείο στο οποίο και λόγω ελλείψεως χρόνου δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε διεξοδικά μεταξύ μας. Θα ήθελα να προξενήσω εγώ ένα διάλογο εδώ. Βεβαίω, θέλουμε να είναι πιο γνωστό το μέσον και έχοντα την πρωτοβουλία να μπορούν να βρουν λύσεις και να βλέπουν κάποιες προτάσεις για την προβολή των προτάσεών τους. Όμως θέλουμε πράγματι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός να διαθέτει κονδύλια στην ε, πρωτοβουλία των πολιτών για προβολή και διαφήμιση της. ξέρουμε πολύ καλά πόσο δαπανηρή είναι η διαφήμιση μέσω του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι και ο τρόπος να καταστεί πιο γνωστή η πρωτοβουλία των πολιτών. Υπάρχουν πολλές και πολυσχεδείς άλλες ε, δυνατότητες. Εγώ θα ζητούσα τουλάχιστον για το σημείο αυτό να γίνει χωριστά η ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα που με ενδιαφέρει είναι, γιατί το συζητήσαμε επί μακρόν, εάν ε, η πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να επιφέρει ε, ή μπορεί να ζητεί τροποποίηση των συνθήκων. Εδώ επικρατούν διαφορετικές απόψεις. Αν κοιτάξουμε όμως το κείμενο, ε, με μία διατύπωση υπάρχουν, υπάρχουν σε ένα σημείο δύο προτάσεις διατύπωση. Στον ΜΠΕ καταρχάς εκεί όπου γίνεται έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει αν μπορεί να τροποποιηθεί το πρωτογενές δίκαιο από, ή να προτείνεται η τροποποίηση πρωτογενούς δικαίου από το Πρωτοβουλία των Πολιτών. Περιμένουμε εν προκειμένου πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ποια θέματα θα μπορούσαν να υπαχθούν στη δυνατότητα αυτή. Εγώ θα πρότεινα να είχαμε σε μια αιτιολογική σκέψη την παρατήρηση ότι θα έπρεπε μια σχετική πρόταση, η οποία θα έχει σε συνέπεια τροποποίηση των συνθηκών, να υπάγεται σε απόφαση, σε προδικαστικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν να εκδώσει απόφαση το δικαστήριο να τοποθετείται για να πει ότι ερμηνεύει το εν λόγω μέσων, την εν λόγω πρόταση για πρωτοβουλία των πολιτών, ότι θα έχει την τάδε τη δίνα συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε αρμοδιότητα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκείνο θα πρέπει να αποφασίζει. Είναι άλλωστε πολύ διαφιλονικόμενο το ζήτημα. Ο κύριος Σοφλίν, ο εισηγητής, έχει κατά, ε, κατά τα άλλα νομίζω ε, λάβει και του αξίζουν τα συγχαρητήριά μας όλων Είδαμε μια σειρά από προτάσεις ε, ώστε η πρωτοβουλία αυτών πολιτών να έρθει πιο κοντά ακόμη στον πολίτη και να γίνει και πιο πρακτικά προσβάσιμη στον πολίτη. Η προθεσμία για τη συλλογή των, των υπογραφών θα πρέπει να αποκοπεί από την ε, αυτόματη αυτή διασύνδεση που έχει με την ε, καταχώρησή της αυτό το δωδεκάμινο για τη συλλογή των πληροφοριών των υπογραφών δεν θα πρέπει να εξαρτάται για την έναρξή του από την καταχώρηση της ε, πρωτοβουλίας. Το δικαίωμα του εκλέγην θα πρέπει να πάει στα 16 χρόνια, πιστεύω, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια μερική καταχώρηση πρωτοβουλία των πολιτών. Συμφωνούμε σε αυτό. Ε, Πολλέ είναι οι προτάσει σας. δεν μπορώ να τι αναπτύξω διεξοδικά όλε, αλλά μια τελευταία παρατήρηση. Εσείς ως γιατί ως μπορείτε να κρίνετε για την τελευταία μου ε, τροπολογία, την 127, εκεί όπου ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει το χέτερο δυνατό τον κανονισμό του σχετικό με την πρωτοβουλία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ καταρχάς να συγχαρώ τον ε, κύριο Σέφλιν ε, για τη δουλειά του και να πω ότι εγώ είμαι ικανοποιημένο ε, με το κείμενο των τροπολογιών συνολικά όπως κατετέθησαν και να πω ότι ο συγκητής έχει λάβει υπόψη τα περισσότερα. Μία αμφιβολία, μία απορία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως και προς ε, τον Γιώργο και τη Σιλβή για ένα θέμα στο οποίο έχω αναφερθεί και συγκεκριμένα πρόκειται για ένα περιορισμό που βάζουμε σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που επηρεάζουν το πρωτογενές ή αφορούν το πρωτογενές δίκαιο αυτές να μην μπορούν να ε, προχωρήσουν. Εμείς στην έκθεσή μας προσπαθούμε να ανοίξουμε λίγο το φάσμα, να διευρύνουμε λίγο το φάσμα ε, στο δίκαιο, σε ό,τι αφορά δηλαδή το δικαίωμα για πρωτοβουλία των πολιτών. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε ε, τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν πιο εύκολα να καταθέτουν περισσότερες πρωτοβουλίες και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές, προπο, ε, πολλές πρωτοβουλίες ε, που μπορούν να κάνουν ε, τον πολίτη να νιώσει Ευρωπαίος και που μπορούν να επηρεάσουν το πρωτογενές δίκαιο. Γνωρίζω πολύ καλό ότι το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί από μία πρωτοβουλία από πολιτών. Απαιτείται ειδική διαδικασία, διότι φυσικά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κατά πάσα πιθανότητα μιας σύμβασης, μιας συνέλευσης ή δεν ξέρω ποιες άλλες διαδικασίες. Όμως ε, το να αποτρέπουμε ή το να απαγορεύουμε ε, πρωτοβουλίες που μπορεί να αφορούν ε, και να επηρεάσουν ένα πρωτογενές δικαίωμα. Και επαναλαμβάνω ότι πολλά, πολλές είναι πρωτοβουλίες που αγγίζουν ακροθυγώς αυτά τα δικαιώματα, το, το, το πρωτογενές δίκαιο, το να τις αποκλείουμε μόνο και μόνο με κριτήριο ότι επηρεάζουν το πρωτογενές δίκαιο, νομίζω ότι είναι υπερβολικό και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έλεγα να μπορεί να υπάρχει μια απάντηση στις ε, προτάσεις αυτές, είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή να εντάσσονται ε, στον προβληματισμό για μια γενικότερη τροποποίηση σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ τώρα Φάμπιο. Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σέφινη εκ πάθους καρδίας για τα, τη δουλειά που έκανε αλλά και για αυτό το πολύ ευχάριστο και άνετο κλίμα μέσα στο οποίο δουλέψαμε στους ε, σκιώδεις. Έγιναν προσπάθειες ε, και για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και καταφέραμε σε αυτό το καλό κλίμα να αντιμετωπίσουμε σειρά προβλημάτων που ε, είχαν δυναμητήσει και την προσπάθεια από πλευρά των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Η μείωση λοιπόν των φραγμών των εμποδίων είναι πρώτος στόχος γιατί διαφορετικά ε, ε, στην ουσία θα, δεν θα είναι δυνατή η πραγματική ε, άσκηση του δικαιώματος των πολιτών. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι οι τροπολογίες J και I, e, e, όπου αναφέρεται ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ε, και όπου από τη μία πλευρά ε, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ε, η αποδοχή της βάσης και από την άλλη πλευρά ε, το ενδεχόμενο από πολιτική άποψη να δοθεί συνέχεια στην ε, πρωτοβουλία, ε, εδώ να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και κατά αυτή την έννοια θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πυροδοτήσει νέες προσπάθειες έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επί της τροπολογίας αυτής με ευχαρίστηση άκουσα ότι θα ξαναγίνει συζήτηση και νομίζω ότι η αξιολόγηση βάσης είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο, ε, η συνάδελφος Κάουφμαν έλεγε προηγουμένως ε, κάτι για τον, ε, την άλλη συμβαστική πρόταση. Καταλαβαίνω τις πρώτες παρατηρήσεις Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα ενδεχομένως να ε, μην χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό για συγκεκριμένους στόχους ή για συγκεκριμένες εκστρατείες, αλλά να προωθηθεί ε, ε, σημαντικά από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, το ίδιο το εργαλείο, έτσι ώστε να καταλάβουν, να το γνωρίσουν οι πολίτες, να καταλάβουν ότι έχουν την δυνατότητα αυτή και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνει πιο προσβάσιμο και πιο εύκολα χρησιμοποιήσιμο. γιατί βλέπουμε ότι και το Ινστιτούτο της Άμεσης Δημοκρατίας έχει πάρει το δρόμο του και θα συμβάλλει και αυτό. Να, για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το εξαίρετο κλίμα που ε, είχαμε στις συζητήσεις και ελπίζω ότι θα εγκριθεί σύντομα και θα προχωρήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Καζιμίρ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέπφλιν και για τη δουλειά του, αλλά και για την κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνει η έκθεση αυτή, ότι είναι σαφές πλέον το περιεχόμενο και ο στόχος που είναι να ενισχυθούν οι θεσμοί, να βελτιωθεί η επικοινωνία και να πάρει περισσότερη υπόσταση αυτή η πρωτοβουλία από ό,τι είχε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να αναπτύσσουμε κάποιους μηχανισμούς ε, που εσωτερικά έχουν παραλύσει. Παρότι μπορεί οι πολίτες ε, να τις έχουν εγκρινεί ή να τις έχουν προωθήσει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να διορθώσει παλαιότερα σφάλματα. Και δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο που ζήτησε να μην ψηφίσουμε ε, τη διάταξη που κάνει λόγο για αλλαγές στον ε, κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Εγώ στηρίζω ακριβώς αυτή τη διάταξη, διότι στη συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί κανείς να ε, φανταστεί διάφορες επιλογές και υποθέσεις. Ο κύριος Σέφλιν ε, με την έκθεσή του μας παροτρύνει εντός του νομικού πλαισίου που καθορίζεται από τις συνθήκες να δώσουμε τα ισιότερα δυνατά εργαλεία σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει πάντοτε να βασιζόμαστε στις ετοιμιγορίες του δικαστηρίου. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, αλλά θα μπορούσαμε και εμείς με δική μας πρωτοβουλία να προχωρήσουμε. Εγώ στηρίζω την έκθεση και τη συμβαστική βή. που ζητάει η Κομισιόν ε, να ξεκινήσει ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ λοιπόν πρόεδρος, ο Μόρτεν Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα για να συγχαρώ τον εισηγητή για το εξαιρετικό αυτό σχέδιο ιδιαίτερα για τα κεφάλαια που αφορούν τις τεχνικές δυσκολίες που είναι τεράστιες και από τα σχόλια που είδαμε και από πολίτες που είχαν εμπλακεί σε αυτές τις ε, προσπάθειες. Στην πολιτική μπορεί να είναι πολύ σύντομος χρόνος το ένα έτος. Ιδιαίτερα αν χρειάζεται κανείς να υπαχθεί σε αυτά τα φορμαλιστικά κριτήρια. Για τους φίλους από τη σοσιαλιστική ομάδα θέλω να επισημάνω ότι δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε στο φάσμα ε, των δραστηριοτήτων σε σχέση με τεχνικά κριτήρια. Αν θα πρέπει δηλαδή ε, μια πρωτοβουλία να επιτρέπεται να αναπτυχθεί ανάλογα με το αν αφορά το πρωτογενές, το δευτερογενές ή το παραγωγό δίκαιο. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση στο να φέρουμε τον πολίτη πιο κοντά και άρα να περιορίσουμε στο δυνατόν περισσότερο τους περιορισμούς. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την εποχή που συντάχθηκε η συνθήκη της Ρώμης. Γιατί λοιπόν να μην μπορούν οι πολίτες να διατυπώσουν μια καλή πρόταση και με ένα εκατομμύριο υπογραφές να την προωθήσουν. Και αν θέλουν ακόμη να αλλάξουν και τη συνθήκη, να ζητούν την αλλαγή τη συνθήκη με ένα εκατομμύριο υπογραφές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τέτοιου περιορισμού. Η πρόεδρος δεν βλέπω να ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Μαϊτέ. Μαϊτέ Ρουίς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σέφλινγκ. Δεν ε, ε, μπορούσε να το κάνει ο ενδιαφερόμενος άμεσα, το κάνω εγώ. Ε, λοιπόν, ε, όσον αφορά τον συμβιβασμό S, λατινικό, όλες οι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών να γίνει πραγματικό εργαλείο, με βρίσκουν σύμφωνοι. Υπάρχουν, υπάρχει όμως κάτι το οποίο κατά την άποψή μας μπαίνει σε, στα όρια της νομικής ασφάλειας, ανα, ασάφειας συγγνώμη, και ανασφάλειας. Ε, αυτός ο στόχος του ενός εκατομμυρίου εάν, εάν ε, ε αναιρεθεί αυτή η βεβαιότητα και πούμε σχεδόν ένα εκατομμύριο, τότε μπαίνουμε σε, στο έδαφος της νομικής αβεβαιότητας. Ή θα είναι ένα εκατομμύριο ή δεν θα είναι. Τα σχεδόν δεν μπορούν να συμβάλλουν στην νομική βεβαιότητα. Όσον αφορά τώρα το ΖΕΝΤΑ, οι ουδέτερες επιτροπές και οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν. Δηλαδή οι ακροάσεις μπορούν να γίνουν είτε από την ΠΕΤ είτε από άλλη επιτροπή. Ε, μια επιτροπή που μπορεί να είναι ουδέτερη μεν, αλλά να γνωρίζει το θέμα ε, για το οποίο συζητάει, ε, το οποίο πραγματεύεται η πρωτοβουλία. Ε, όσον αφορά το λατινικό γιου είναι μπερδεμένο το θέμα. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει το εργαλείο, θέλουμε να έχουν αυτή τη διευκόλυνση οι πολίτες, αλλά η δημόσια χρηματοδότηση ε, περιλαμβάνει κινδύνους κατά την άποψή μας, ε, κινδύνους ε, όσον αφορά χρήσεις που δεν θα είναι αυτές που πρέπει ή ότι θα ξεκινήσουν ενδεχομένως κάποιοι κάποιες πρωτοβουλίες για να αυτοχρηματοδοτηθούν κτλ ενδεχομένως θα πρέπει με άλλο τρόπο να βρούμε, να βοηθήσουμε ε, τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Δεν ε, συμφωνώ με την εξάντε, με την εκ των προτέρων δημόσια χρηματοδότηση εξπόστ, ναι. Thank you very much. I, don't know, George, if like to, to respond. Ευχαριστώ, George. Α, δεν είδα, δεν είδα Έχω όλη τη γραμματεία εδώ δίπλα μου, αλλά κανείς δεν σας είδε να σηκώνετε το χέρι σας. Δεν σας, δεν σας είδαμε, κύριε Τερικάμπρας. Και μάλιστα δεν σας είχα δει να θέλετε να μιλήσετε και εξεπλάγει. Visibility back. Thank you very much. Θα απαιτώ να ξανακερδίσω την ορατότητά μου, να με βλέπετε. Τρία σημεία. Well, in, paragraph, in par, ε, ε, just excuse me. The, the question, the question of the of the mother tongue, uh, which uh, Sylvie Kaufman treated, I think. Το θέμα της μητρικής γλώσσας. Θα ήθελα να ξέρω γιατί ο αγαπητός κύριος Σέφλινγκ δεν έλαβε υπόψη όλες ε, τις τροπολογίες. Η τροπολογία μου 21 νομίζω ότι εν μέρη θα μπορούσε να ε, λύσει το ζήτημα. Δεύτερον, συμβιβαστική S. Πούντο όμως δεν το βρίσκω λέει ο μιλητής. δεν νομίζω ότι τελικά ε, το λύσαμε επιτυχώς. Λέτε ότι σε 12 μήνους, ε, μήνες μετά την ε, σχετική γνωμοδότηση. Τι σημαίνει positive opinion, θετική γνωμοδότηση, ότι έχει γίνει ήδη δεκτό το θέμα ή ότι έχει κριθεί με θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Επίσης, ε, στην ίδια συμβαστική, S ε, αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προτείνει με έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Εδώ έγινε συζήτηση εάν θα γίνει η ίδια πρωτοβουλία ή αν θα είναι η ενέλη έκθεση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πριν φτάσουμε σε συμφωνία επ' αυτού. Τελευταίο σημείο. Συμφωνώ απολύτως με τον φίλο μου Ραμόν Χάουγκη, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει με ένα σημείο που είναι δύσκολο και που αφορά το πρωτογενές δίκαιο. Ωστόσο, άποψή μου είναι ότι ο Σάρφος Κάουφμαν έκανε κάτι σωστό. Εν μέρη, εν πάση Εν μέρη, εν μέρη. Δηλαδή, η Κομισιόν δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει το δικαστήριο. Η Κομισιόν όμως μπορεί να, να πει να να, έχει πολιτικό λόγο. Ε, ο νομικός λόγος θα βαραίνει το δικαστήριο. Και επομένως όσο περιμένουμε τον νομικό λόγο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τον πολιτικό λόγο. Δηλαδή ποια είναι η άποψη της Κομισιόν από αυτού. Αυτή είναι η άποψη. My grateful thanks να ευχαριστήσω τις ευχαριστήσεις μου σε όλους για τα σχόλιά τους που είναι άκρος πολύτιμα. Και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω όλα αυτά στο τελευταίο κείμενο που έχουμε σας παρουσιάσει και το οποίο ελπίζω να είναι έτοιμο αύριο. Συγκεκριμένο τώρα να κάνω κάποια σχόλια. Πράγματι το θέμα της γλώσσας ε, διχάζει τις διάφορες ομάδες. Αναγνωρίζω το γεγονός αυτό. Προσωπικά θα έκλεινα να είναι ευρύτερο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ζήτημα κόστος και άλλα ζητήματα, αλλά επί της αρχής λέω ότι περίπου το 10% ε, των πολιτών της Ένωσης δεν μιλάνε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα ήταν δίκαιο να τους αποκλείσουμε. Τη διατύπωση την επεξεργάζομαι και με λίγη τύχη ελπίζω να βρω μια διατύπωση που θα σας ικανοποιεί όλους, αλλιώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν τμήματικές ψηφοφορίες, έτσι είναι η ζωή όμως, τι να κάνουμε. Τώρα να προχωρήσω. Α, ναι. Με την πρωτογενή νομοθεσία αυτό το πρόβλημα. Αυτό που λέει ο Ραμόν Χάουριγκ είναι πολύ ενδιαφέρον θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ένας τρόπος αποθήκευσης των ε, εν λόγω πρωτοβουλειών. Πρέπει να το σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει. Μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Ε, δεν μπορεί μια πρωτοβουλία να τροποποιεί το πρώτο δίκαιο, αλλά είναι ένα πολύτιμο σχόλιο που μπορούμε να το ε, λάβουμε υπόψη και το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι. Μάλιστα. Α, αυτό πάει σε αυτά που είπε η Μάιτε. Ναι, θα δω να βρω, ε, θα δω μπορώ να βρω τη διατύπωση που θα είναι καταλληλότερη. Πάντως δυσκολεύομαι με αυτό που λέτε ε, για την Επιτροπή ε, οι πιο πολλοί πολίτες ε, δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Μια επιτροπή δηλαδή που επηρεάζεται να είναι μια επιτροπή με την οποία έχουν κάποια επαφή. Γιατί δεν τους αρέσει. Φυσικά θα είναι αρνητική μια τέτοια επιτροπή να επηρεάζεται. Εμείς θα έπρεπε νομίζω να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα διεξάγουμε τις ακροάσεις αυτές. Αυτό που είπατε για τη δημόσια δαπάνη, η κυρία Κάφμαν για την τηλεόραση, ξέρετε η τηλεόραση είναι ακριβή. Τα ραδιόφωνο όχι. Για τον κύριο Τερικάμπρας. Νομίζω ότι είναι και νομικό και πολιτικό ε, αυτό το έργο της, Κομισιό, της Επιτροπής. Και φυσικά το δικαστήριο του Λουξεμβούργου είναι από τη νομική αρχή, αλλά για την πολιτική αρχή ποιοι είμαστε εμείς, είναι το κοινοβούλιο. Δεν είναι σαφές. Και αυτό έχει και να κάνει με το πώς λειτουργεί ως πολιτική οντότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Αν την ξέρετε εσείς παρακαλώ μέσω γραπτής διαδικασίας να με ενημερώσετε και εμένα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε λοιπόν θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στις 28 του μήνα την έκθεση και μάλλον στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Θα πάει στην Ολομέλεια. Πηγαίνουμε στο επόμενο σημείο που είναι η γνωμοδότηση του Πάλο Ρανζέλ γνωμοδότηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο Πάουλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να πω ότι δυστυχώς δεν θα είμαι παρόν στην ψηφοφορία της απόμας γιατί έχουμε εκλογές όπως ξέρετε στην Πορτογαλία στις 4 Οκτωβρίου άρα την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη τουλάχιστον θα πρέπει να είμαι στην περιφέρεια για την προεκλογική εκστρατεία. Και τώρα να συνεχίσω στα πορτογαλικά για να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης. Η πρόεδρος, παρακαλώ, λίγο πιο σιγά. Λοιπόν, σχέδιο γνωμοδότησης για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αθμιστικών οργάνων και φορέων και μάλιστα διεθνών οικονομικών ομισματικών επίσης οργάνων και οργανισμού. Η οικονομική διακυβέρνηση γίνεται σε φόρουμ όπως είναι ο ΣΑ, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ομάδα των 20, η Επιτροπή της Βασιλείας, FSB, πρόκειται για φορείς, για οργανισμούς πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους Όμως, είναι και τελείως διαφορετικό το επίπεδο, το θεσμικό του καθενός. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιους ε, διεθνείς χρηματοδοτικούς καθαρούς, αμυγός χρηματοδοτικούς όπως είναι το ΔΕΛΤΑ αλλά έχουμε την ομάδα των 20 για παράδειγμα, που είναι κάτι πιο άτυπο. Ή έχουμε τα λογιστικά πρότυπα και τους οργανισμούς σχετικούς άλλους δηλαδή πιο ιδιωτικούς φορείς επίσης, Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι πιο σημαντικέ από αυτούς, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους ε, διεθνείς χρηματοπιστωτικού φορείς. Εγώ προσπαθώ να δω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών και τι καθεστώς έχει σε κάθε έναν από αυτούς τους οργανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, προσπαθώ να δω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τη βελτιστοποιήσουμε. Θα τόνιζα λοιπόν εδώ ότι αν εξετάσουμε τους ε, οργανισμούς αυτούς θα δούμε ότι είναι ετερόκλητοι, είναι τελείως διαφορετικοί ε, το G20 για παράδειγμα. Είναι μια, ε, μια συνέλευση λήψης πολιτικών αποφάσεων, άτυπη όμως. Ένα φόρουμ κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι θεσμικός ο χαρακτήρας. Αν συγκρίνουμε ε, το G20 με τον Διεθνές Μεσοδοτικό Ταμείο, βλέπουμε τις διαφορές. Είναι θεσμοθετημένο και έχει ένα πολύ έτσι παγιωμένο θεσμικό χαρακτήρα εδώ και χρόνια το ΔΝΤ. Έχουμε λοιπόν κάποιες ανησυχίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, τι ε, πώς μπορεί να επηρεάσει, πώς επηρεάζει και αν επηρεάζει αυτά τα όργανα τους οργανισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την περίπτωση του g Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται θεσμικώς από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Εκπροσωπούνται όμως και ορισμένα από τα κράτη-μέλη. Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Και στην περίπτωση τώρα του ΔΕΛΤΑ και του ΩΣΑ, εκεί εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν όλοι. Γιατί δεν είναι στον ΩΣΑ. όχι, στο Διεθνές Ταμείο δεν είναι όλα. Ε, Εκεί έχει καθεστώς παρατηρητή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές ε, συνεδρίες οι οποίες ε, παρίστανται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συστηματικά, δεν είναι θεσμοθετημένος ο ρόλο τη Ένωση. Ε, υπάρχει κάποια αταξία, θα έλεγα. Δεν υπάρχει μια συνεκτικότητα της παρουσίας και του καθεστώτος της Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλου αυτού του φορεί και όργανα. Και αυτό επαναλαμβάνω γιατί είναι τελείως ατερόκλητοι μεταξύ τους και οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί. Άρα απαιτείται διαφορετικού είδους εκπροσώπηση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό είναι το ζήτημα του δημοκρατικού ελέγχου. Το accountability όπως το λέμε, ε, την ε, υποχρέωση λογοδοσίας. Και εδώ είναι το θέμα της εκπροσώπησης πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει πολλές ανταλλαγές απόψεων για το θέμα και το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε αρκετές φορές. Πιστεύω όμως ότι καλό θα ήταν, για παράδειγμα, να έχουμε πριν από τις συνεδριάσεις ε, της G20 ένα διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον πρόκειται να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις παγκόσμιου βεληνικούς που επηρεάζουν και την ευρωπαϊκή ε, θέση, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων πριν από τις συνεδριάσεις ε, του G20. Και το ίδιο να γίνεται και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν χώρες, παρεμβαίνουν, έχουμε και την Τρόικα και ε, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές μεταξύ των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δούνου Αυτό θα αιτιολογούσε και τη δική μας παρουσία και τη δική μας συμμετοχή, να είναι ευρωπαϊκή η συμμετοχή και όχι η συμμετοχή να είναι μεμονωμένα των κρατών μελών. Και ένα τελευταίο τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνεια σε αυτόν τον οργανισμό και εξηγούμε. Αυτά τα θεσμικά, μάλλον αυτά τα όργανα έχουν ε, τεχνική φύσεω ε, έργο. Για παράδειγμα, η Επιτροπή τη Βασιλεία, οι έργοι που ρυθμίζουν τα ε, αξιόγραφα ε, με τι τράπεζε. Έχουμε και την περίπτωση ενό ταμείου που θεωρήθηκε ω μαύρο ταμείο μια τράπεζα. Υπάρχει έλλειψη διαφάνεια. Υπάρχει ένα είδο αδιαφάνειας, έλλειψης ορατότητας και πολλές φορές πίσω από τα άκρος τεχνικά ζητήματα συγκαλύπτονται, κρύβονται πολύ λεπτά πολιτικά ζητήματα. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραλαμβάνω, πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις ε, οργανώσεις. Ε, είμαστε μέλη, αλλά προς του Συμβουλίου και της Κομισιόν και οι δύο προσωπούν και πρέπει να εκπροσωπούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ένωση και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πλήρες μέλος ε, και του ΩΣΑ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί σε άλλους οργανισμούς πιο ιδιωτικού χαρακτήρα, δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν αποδεκτό ε, ο καθώς παρατηρητή, αλλά σε κλασικούς οργανισμούς, αν σου προανέφερα, θα ήταν ενδιαφέρον. θα μπορούσε να πει κανεί ότι στο δούνο του εκπροσωπούνται κάποια κράτη. Ναι, είναι σαφέ. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα γενικό ενδιαφέρον ευρωπαϊκό και μετά να υπάρχουν περιπτώσεις όπως η πολύ κραυγαλαία περίπτωση του G20 όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταφέρει τι θέσει και, και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα όχι μόνο των εκπροσωπούμενων σε τη χώρο, αλλά και των χωρών και θα έλεγα περισσότερο ε, μάλλον ακόμη αυτών των χώρων που δεν εκπροσωπούνται εκεί. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχει καθεστώ ε, μόνο παρατηρητή στο Νοσά, επαναλαμβάνω, και, στη, και στο Δεύτερο Μεσοδοτικό Ταμείο η Ένωση. Αυτό είναι το δεύτερο. Δεν έχει να κάνει με το καθατικό αυτό, είναι θέμα μεθοδολογικό. Πρέπει να έχουμε έναν τρόπο δουλειάς, μια μέθοδο εργασίας για να υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές που λαμβάνονται στα φόρα αυτά. Γι' αυτό και θα πρέπει να μπορούμε να εκπονούμε κοινέ θέσεις. Και αυτό σχετίζεται με τη διαφάνεια και τη δημοκρατική ευθύνη, που είναι το τρίτο που ανέφερα. Δεν νομίζω θα ήταν καθόλου άσκοπο ή παράλογο να έχουμε ανταλλαγές απόψεων εκ των προτέρων για να ορίζουμε τις εντολές σε θέματα όπου θα μπορούσαμε να έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα. Ιδίω αν θα εκπροσωπηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις. Και θα πρέπει να γίνει ε, συσχέτιση εδώ και με την εμβάθυνση της ε, Οικονομικής και Νοσηματικής Ένωσης. Έχουμε την έκθεση Μπρόκ Έχουμε και την Εξφερχόφστατ και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, τέλος πάντων ίσως της Ευρωζώνης μόνο. Τουλάχιστον οι χώρες Ευρωζώνης που έχουν κοινά συμφέροντα θα έπρεπε να έχουν μία και μόνη ε, θέση σε, αυτές τις, ε, σε, αυτού, σε αυτούς τους οργανισμούς και φορείς. Και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ κατά την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Άλλες αρμοδιότητες έχει η Ένωση, άλλες τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε την κατανομή. Τώρα, νομιμοποίηση, δημοκρατική ευθύνη, λογοδοσία κτλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι πρέπει να είναι ενήμερο για τη δράση των ε, οργανισμών και φορέων αυτών, να έχει πρόσβαση δηλαδή στα έγγραφα, αλλά να έχει πρόσβαση και στις αποφάσεις. Και αν χρειάζεται, να έχει και αυτές τις ανταλλαγές απόψεων προκαταβολικά για να μπορέσει πριν, παραδείγματος χάρη από μια διάσκεψη κορυφή τη ομάδα ε, των 20, να μπορεί να έχει καταγράψει τη θέση του, να έχει καταλήξει σε μια θέση ώστε να μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη συνέχεια. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιατί? Αφενός γιατί εγγυώνται ότι έχουμε περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, άρα μειώνεται το δημοκρατικό έλλειμμα και απ' την άλλη ε, αυξάνουν και τη διαφάνεια, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι οργανισμοί, ιδίως οι πιο τεχνικοί, είναι και κάπως αδιαφανείς. Επομένως, η συζήτηση σε ένα φόρο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βελτιώσει την κατάσταση αυτή, θα αυξήσει τη διαφάνεια. Υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο, μια τελευταία σύσταση, η τελευταία που θέλω να σχολιάσω. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλει με ηγετικό και πιο ενεργό ρόλο στη μεταρρύθμιση αυτών των οργανισμών. Εμείς λέμε τώρα ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση. Ε, το έχουμε καταλάβει αυτό. Άρα τώρα πρέπει να δούμε και ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι κανόνες και οι τρόποι και της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό θα μπορούσε να στεπάγεται μια μεταρρύθμιση. Πολλές φορές γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑ, το έχουμε ακούσει και ξανακούσει. Έχουμε ακούσει να γίνεται λόγος και για τη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών οργανισμών που έχουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης και ακριβώς εδώ έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει το ρόλο της ε, με τολμηρές ε, τοποθετήσεις, ε, με δυνατότητα πρωτοβουλίας για να προτείνει μεταρρυθμίσεις της παγκόσμια της διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτές είναι οι προτάσεις μου, τόσο ώστε να μπορούμε να προτείνουμε και νέα μοντέλα και βέβαια η συμμετοχή στους διεθνούς οργανισμούς ε, και φορείς. Ε, έχουμε και την έκθεση Γκουλάρ βέβαια που μιλά για τη ε, συμμετοχή στους οργανισμούς αυτούς της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής κοινωνικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε μία σύσταση γιατί μέρος των προβλημάτων που έχουμε όπως φαίνεται και από την γνωμοδότηση και από την έκθεση, έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτή τη διαφορά που υπάρχει ε, μεταξύ των ε, διαφορετικών αυτών ε, οργανισμών. Και κατά σιγά σιγά. Δεν είναι συγκεκριμένα πολύ ίσως ε, ουσιώδες το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προκύψει από μια γνωμοδότηση, μια έκθεση σαν και αυτή, ακριβώς γιατί έχουμε πολλούς ετερόκλητους οργανισμούς και φορείς για τους οποίους μιλάμε εδώ. Θα μπορούσε όμως γενικά να ενισχυθεί το καθεστώς της Ένωσης και να βελτιωθεί ο συντονισμός μας. Να έχουμε δηλαδή μια κοινή θέση στο πλαίσιο αυτών των διαφόρων φορέων και οργανισμών. Επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ευαισθησία και κοινοποίηση των ε, εκτενόμενων στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών και τρίτον έλεγχος, δημοκρατικός έλεγχος. Με βάση λοιπόν αυτές τις αρχές και με την παρότριση αυτή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στη μεταρρύθμιση των διεθνών αυτών ε, οικονομικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών για να έχουμε μια πιο συνεκτική, μια πιο συνεπή διεθνή διακυβέρνηση με εκπροσώπηση των κρατών με πιο μεγενή τρόπο είναι οι προτάσεις μου. Δηλαδή να προτείνουμε διάφορα μοντέλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αυτή η οποία θα δώσει την όθηση για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι οι τρεις αρχές λοιπόν και αυτές είναι οι συστάσεις που περιέλαβα στην νομοδότησή μου μια γνωμοδότηση που είναι σημαντική. Και ε, να τονίσω ότι ήταν και δύσκολο να καταλήξω γιατί ήταν τελείως ετερόκλητοι αυτοί οι οργανισμοί για τους οποίους έπρεπε να γνωμοδοτήσω. Ευχαριστώ. Ένας μόνος συνάδελφος, ο κύριος Σαουράκη θέλει το λόγο. Κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι για την έκθεσή του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά του και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδίω για τις πληροφορίε που μας ε, δίνει. Δεν το έχω συγκεκριμενοποιήσει ακριβώ, αλλά θα ήθελα να πω ότι πράγματι είναι σκόπιμο και σωστό να είμαστε μέλος στους ε, Διεθνείς Οργανισμούς Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Διαχείρισης. Πρέπει να έχουν την άποψη ότι στην Ένωση γίνονται προσπάθειες οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις ε, να ε, ενταχθούν ε, σε αυτή την προσπάθεια για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται και από του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η Ευρώπη έχει ταυτότητα, θα έλεγα, στο θέμα αυτό. Στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε γίνεται προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση να προωθηθεί η έννοια μιας υπεύθυνης επιχείρησης με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Δεν θα προχωρήσουν αυτά όμως αν οι διεθνείς οργανισμοί G20, Δουνουτού, Ηνωμένα Έθνη και άλλοι που έχουν ε, ιστορικό, ε, που έχουν προϊστορία και μεγάλες επιχειρήσεις ε, Έχουμε την ιδέα, για παράδειγμα, ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν εμπειρία και πρέπει να. Ε, πω ότι έχει δίκιο ο Παύλο που λέει ότι πρέπει να βάλουμε αυτό ε, το ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό Δηλαδή να προωθήσουμε ότι και τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, είναι και σημαντικός φορέας κοινωνικής ε, συνοχής. Και αυτή την δική μας τη στάση θα πρέπει να την ενστερνιστούν και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές Θα προβώ στη διατύπωση μια τροπολογία και ελπίζω να μπορέσει ο να την συμπεριλάβει στο κείμενό του. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλάρ. Όχι, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και όλους διετυπωσαν τύπωσαν σχόλια, μια-δυο διευκρινήσεις μόνο. Πρώτον, έχω αντίληψη όμως ότι υπάρχει ένα τεράστιο εγχείρημα και λύση δεν έχω έτοιμη να προσφέρω. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να δραματίσει χρήσιμο ρόλο, εξασφαλίζοντα την συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος, ε, τη ιστορική διαστρωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων οργανισμών που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε πρόσκεντες επιχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι το ένα. Και επίσης, λογοδοσία, διαφάνεια και ε, παγρύπνηση ώστε να τηρούνται από τους εταίρους μας στην ε, διεθνή κοινότητα οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Αυτό το κάνουμε και εμείς, πρέπει να το πράττουν και εκείνοι. Είναι περίπλοκη κατάσταση, δεν είναι πάντα ε, οι ίδιοι εταίροι και συμπεριφορά τους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να είμαστε αφελείς. να συνεργαζόμαστε δηλαδή σε πολυμερές επίπεδο, αλλά χωρίς να είμαστε αφελείς. Και πρέπει επίσης να δούμε εάν οι διεθνείς κανόνες που επιβάλλονται σε ορισμένους κανόνες, σε ορισμένους ε, τομείς, ε, καταβροχθίζουν το τραπεζικό μας τομέα. Να μην κλείνουμε τα μάτια πρέπει να έχουμε στρατηγική, γιατί έχει στρατηγική, σημασία για την επένδυση στο μέλλον, για τη χρηματοδότηση του μέλλοντος, της ανάπτυξης και των θεσμών εργασία για την Ευρώπη ο τραπεζικός τομέας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και εγώ στη διάθεση του εισηγητή και της χρωματεία μας και της Επιτροπής μας ε, για το θέμα αυτό το δύσκολο, αλλά ένα θέμα που κατεξοχήν και μετά την κρίση μπορεί να, κάνει, να δώσει τον πολίτη να καταλάβει τι προσθέμενη αξία μπορεί να έχει η Ευρώπη σε σχέση με επιμέρους προγράμματα, με επιμέρους ε, προσπάθειες των κρατών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εάν δεν έχετε τίποτα να πείτε. Αν έχετε κάτι άλλο, λοιπόν, για τα δεούς εθνείς ε, οργανισμούς, που πολλές φορές είναι και ανεξάρτητοι, ιδιωτικοί, τα θέματα της λογοδοσίας, ε, όλα αυτά θα τα λάβετε υπόψη λοιπόν και για να καλύψει τον ρόλο της Ένωσης σε αυτό και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ε, φορέων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που πρέπει να είναι ανεξάρτητα, ταυτόχρονα πρέπει να διαφυλάσσουν την αυτονομία τους και να λειτουργούν μέσα σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο αυτά τα δεδομένα. Και άλλη μια ερώτηση που συχνά νομίζω ανακύπτει. Ότι η Επιτροπή που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση διεθνή θεσμικά όργανα. Ε, πώς μπορεί να εκπροσωπήσει την, Ευρωπαϊ... την ΟΝΕ όταν ε, η ΟΝΕ βρίσκεται ακόμη σε διακυβερνητικό ε, επίπεδο. Απάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλες τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους. Για το συνάδελφο Χαουρέχη θα ήθελα να πω ότι βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και υποστηρίζουμε την ιδέα της αηφορίας ιδιωσιμότητας, όχι μόνο σε περιβαλλοντικούς όρους. αλλά και ως κοινωνική διάσταση η προϋπόθεση. Δεν όμως αυτός νομίζω ο στόχος της έκθεσης που έχει θεσμικό χαρακτήρα. Δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θέλουμε να υλοποιήσουμε δηλαδή. Βεβαίω κατά κάποιον τρόπο ε, θα λάβουμε ή θα εισαγάγουμε, θα ενσωματώσουμε την ιδέα αυτή. Αλλά βασικά η ιδέα είναι να καλύψουμε τα θεσμικά ζητήματα που υπάρχουν εδώ. Για τη Σίλβι Γκουλάρ, η για την ΕΚΟΝ. Συμφωνώ κατ' ουσίαν με τις ιδέες που έχει αναπτύξει και πρέπει να πω ότι το γεγονός και μόνο που μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι η διάγνωση αυτή τη στιγμή και δεν συμφωνώ. Αλλά πάντως το να μπορούμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα που δίνει αυτή η κατάσταση. Το να αντιληφθούμε ότι υπάρχει πραγματική διαφορά μεταξύ της Επιτροπής της Βασιλείας και του Ιδουνοτού ή της χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης ε, και του G20. Ήδη αυτό σημαίνει και διαφορετική, διαφορετικό τύπο εκπροσώπηση αλλά και διαφορετικό είδος λογοδοσίας. Και άρα είναι ήδη αυτή η πηλιά πάρα πολύ χρήσιμη. Διότι μέχρι τώρα ήταν θέματα τελείως χωριστά αυτά. Και έτσι φτάνουμε στην πρόταση που διατυπώνεις ότι μπορεί να διαμορφώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση έτσι ώστε να εκπροσωπούνται κάποιοι θεσμοί τουλάχιστον και έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία με διαφορετικούς φορείς και θεσμικά όργανα και έτσι μπορούμε να τα υπαγάγουμε σε μια ομπρέλα ε, όπου θα εκπροσωπούνται. Βέβαια τα πιο δύσκολα ερωτήματα τα διατυπώνει η Πρόεδρος, πρέπει να πω. Γιατί το δύσκολο είναι να γνωρίζουμε, επί παραδείγματι, αν θα πρέπει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να διαδραματίζει ρόλο. Σε καθαρά οικονομικά ζητήματα, κατά πάσα πιθανότητα όχι, αλλά πάντως ε, σε σχέση με τους μόνιμους εκπροσώπους και το ρόλο τους μπορεί να διαδραματίζει ρόλο. Και νομίζω ότι υπάρχει όντω η δυνατότητα και είναι σαφέ σε ορισμένε περιπτώσει ότι θα πρέπει η ΕΚΤ να είναι παρούσα και στους φορείς και τα θεσμικά όργανα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και κατά πάσα πιθανότητα σε αποφάσεις του G20. Με τι καθεστώς όμως, γιατί εδώ πρόκειται για ένα φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεν ανεξάρτητο δε. Και άρα είναι δύσκολη η διαχείριση του θέματος. Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να το δούμε για τη συνεργασία μας ως εμπειρογνωμόνων μπορεί ίσως να είναι πιο ευεπίλητη γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει. Με συγχωρείτε, σαν το κινητό μου. Μπορεί να ε, λύνεται λοιπόν σχετικά εύκολα, αλλά υπάρχουν και άλλες δυσκολίες εδώ. Έχουμε λοιπόν ε, φτιάξει ένα μόρφωμα μάλλον αφηρημένο, γιατί δεν λύνει όλα τα ζητήματα. Και είναι άλλο πράγμα να δούμε τις ε, θέσεις μας στην στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς και να τους διακρίνουμε από άλλα όργανα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν τη διαφοροποίηση. Δεν πρέπει όμως να προκαταλαμβάνουμε την όποια απόφαση πρόκειται να δοθεί. Με διαπραγμάτευση πιστεύω, όταν διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και πάντα στο πλαίσιο των συνθήκων ε, που θα τροποποιηθούν έτσι, που διαμορφωθούν έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εκπροσώπησή μας στους διεθνείς φορείς και αντίστοιχα πρέπει να διαμορφωθούν οι λύσεις και για την Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν στο στάδιο αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση στα ζητήματα αυτά. Βεβαίω, εάν γίνει η μεταρρύθμιση της ε, ε, παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, ασφαλώς θα είναι ε, πιο εύκολο να πείσουμε τους διεθνεί οργανισμού για αυτό το νέο θεσμικό σχεδιασμό. Αλλά μέχρι τότε εγώ μάλλον θα προτιμούσα να εμείνω στη βασική αρχή, δηλαδή να είμαστε και μέλη του Διοδούνου του και του ΟΣΑ και να μπορούμε να συντονίζουμε κοινέ θέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κέντρα αυτά και και αυτό νομίζω πρέπει να αναπτύξουμε ως ε, επιδίωξη, να συζητήσουμε λεπτομερέστερα και να, συζη... και να προσκαλέσουμε τους διάφορους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών αυτών φορέων να έρθουν στην ε, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, την Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων, να προβούν σε συνομιλίες με τους βουλευτές πριν αλλά και μετά από κάποιες καθοριστικές αποφάσεις και συναντήσεις για να συστήσουμε μαζί τους και να συζητήσουμε και τι είδους εκπροσώπης θέλουμε. για να συζητήσουμε το θέμα της εκπροσώπησης και της νομοποίησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκείνο βέβαια το οποίο ιδιαίτερα απασχολεί πολλούς και προκύπτει ο ζήτημα κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε ε, για διάφορες πολιτικές ε, και άλλες ε, περιπλοκές που είναι το ζήτημα της διαφάνειας διότι κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας αλλά και άλλοι το τρόποι η τεχνική που υπάρχει για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των ισολογισμών των εταιριών λοιπά Έχουν, κρύβουν πίσω τους πολιτικές, ε, πολιτικές συλλογιστικές περίπλοκες και που θα πρέπει να εξετάσουμε βεβαίως και με βάση και τις ευθυντήριες γραμμές που προσδιορίσαν τα αρμόδια πολιτικά όργανα. Άρα τα ζητήματα της διαφάνειας μπορούμε να τα βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όπως είπα θεωρώ ότι οι δικές σας ερωτήσεις, αυτές ιδιαιτέρες που αφορούν το ποιος και με ποιο ρόλο. Θα εξασφαλίσει και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και την παρουσία της ορισμένου φορεί. είναι πράγματι πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά όπως έχω ήδη πει είναι πολύ πρόωρο το να δώσουμε απάντηση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν μπορεί να πάρει το λόγο εάν ενδιαφέρεται. Αν δεν θέλετε δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλώς σας δίνω την ευκαιρία να μας επικρίνετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εγώ προέρχομαι από την Γενική Διεύθυνση Εκφίνα. και η Γενική Διεύθυνση 20 επίσης ε, ασχολείται με αυτά τα θέματα εν μέρη. Αυτό που είπε η κυρία Γκουλάρη είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα που καλά το είπε. Πρόκειται για χαρτογράφητα ύδατα. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να είμαστε μέλη του ε, Διεθνούς Ομοσματικού Ταμείου ε, και τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ε, θα πρέπει, εάν ε, γίνει, να γίνει με υποστήριξη του 85% των ε, μέτρων. Όσον αφορά τώρα αυτά που αναφέρατε, όσον αφορά ε, την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ε, την ενωσιακή προσέγγιση όπως την αναφέρατε. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Ο πρόεδρος μας έχει δεσμευτεί να υποβάλει γρήγορα ε, πρόταση την οποία θα υποβάλει και στο Ευθύνες Νομισματικό Ταμείο και μάλιστα το ανέφερε και στο, στην ομιλία του ενώπιου του Κοινοβουλίου για την, ε, για την κατάσταση της ε, ενώσεως. Δεν ξέρουμε πότε η πρόταση θα υλοποιηθεί, πάντως σύντομα Ωστόσο, είναι σαφές ότι η, ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι καλοδεχούμενος ε, ε, και η συμβολή του στο θέμα αυτό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ υπάρχει μία πρόνοια η οποία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς αλλά σεβόμενοι το άρθρο 138 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε αποφασιστεί ε, μετά από πρόταση της Κομισιόν, ε, οτιδήποτε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, θα αναφέρεται οπωσδήποτε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Thank you ε, very much. <clears throat> Πολλές οι προκλήσεις, πολλά τα θέματα αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε προχωρούμε προς την ε, συνολική διακυβέρνηση και θα πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι καταλήλως. Έστω και αν σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε τελικές λύσεις, ε, εκτιμούμε την εργασία της ε, Σιλβή και βεβαίως του συντάκτη μας. Να σας πω ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στις 22 Οκτωβρίου θα συζητηθούν ε, οι τροπολογίες. Αυτά λοιπόν και ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ξαναρχίσουμε αύριο στις 10, αλλά θα παρακαλέσω τους συντονιστές να παραμείνουν γιατί...